Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να καθίσετε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ε, Περιφερειών, εξ Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εξ αρχής θα ήθελα να δώσω το λόγο στους διερμηνείς μας που είναι ε, πολύ ευγενική μαζί μας και σήμερα θα δουλέψουμε όλη την ε, ημέρα, αλλά μου ζήτησαν να μπορέσουν να διαβάσουν ένα σύντομο μήνυμα ε, για να μας εξηγήσουν τι συμβαίνει. Ε, από τους διερμηνείς σας λοιπόν να σας πούμε ότι βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω της εργασιακής διάνεξης με τη διοίκηση για τις συνθήκες εργασίας μας. Σε ορισμένες καμπίνες έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διερμηνείς και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Αυτό ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμά μας στην απεργία και συνιστά διάκριση προς τις υπόλοιπες γλώσσες. Ω εκ τούτου και σε ένδειξη αλληλεγγύη, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει στη στάση εργασία που προβλεπόταν για τη σημερινή συνεδρίαση και η συνεδρία θα τελειώσει στην προβλεπόμενη ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ήταν ένα σύντομο μήνυμα από τους διερμηνείς, τους οποίους εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τη σπουδαία δουλειά που κάνουν για μας και θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε ακριβώς στις 12.30. Θα είναι πιο εύκολο για μας. Ε, ε, ξεκινάμε τώρα τη συνεδρίασή μας, 20 ε, ε, Απριλίου σήμερα, όλη μέρα έχουμε συνεδρίαση, θα έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη, συμφωνείτε για την ημερήσια διάταξη αυτή. Μάλιστα, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Ε, από προηγούμενες συνεδριάσεις λοιπόν έχουμε τα πρακτικά, είναι διαθέσιμα επιγραμμικά, online, μπορείτε να τα δείτε, να τα μελετήσετε και όσοι ήθιστε, εάν δεν υπάρξουν ε, ενστάσεις μέχρι το τέλος της σημερινή συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι γκρίνονται. Τρίτο σημείο, ανακοινώσεις της Προέδρου. Με χαρά σας ανανημερώνω ότι τις ε, περασμένες εβδομάδες είχαμε δραστηριοποιηθεί ε, ως εκπρόσωποι της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συμμετείχαμε σε διάφορες σημαντικές συνεδριάσεις. Στις 7 Ιουνίου έγινε μια συνεδρίαση στην Επιτροπή των Περιφερειών όπου συμμετείχε ο κύριος Φανίστελ Ρόι ε, ως ομιλητής και εγώ. Παρουσιάσαμε τη θέση της Επιτροπής Ρέτζη για την πολιτική συνοχή και για το μελλοντικό PDP. Παρακολουθήσαμε αυστηρά την έκθεση της Επιτροπής Περιφερικής Ανάπτυξης και τη θέση μας, καθώς και τις συστάσεις που είχαμε ειδικά την έκθεση του κύριου Ρουγούα για την ε, ε, έκθεση της Επιτροπής και ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου αναπτύξαμε τη θέση της Επιτροπής μας. Στις 8 ε, ε, Ιουνίου διοργανώθηκε ενδιαφέρουσα συνεδρίαση από τη Βουλγαρική Προεδρία και εκεί ε, Είχαμε μια παρουσίαση της Αναπτυξιακής Επιτροπής. Η κυρία Βέστφαλ ήταν η ομιλήτρια και συμμετείχε. Ο κ. Βανίς Ρόιτ επίσης. Οπότε, τρεις εξημών παρουσιάσαμε τη θέση της Επιτροπής μας και συμμετείχαμε στη συζήτηση και έπειτα μιλήσαμε για τη θέση αρκετών κρατών μελών σε σχέση με τη μελλοντική πελωτική συνοχή. Ήταν λογικό να παρουσιάσουμε τη θέση της Επιτροπής μας ως θέση του Κοινοβούλιου, γιατί υπογράμμισα κιόλα στη διάρκεια της των εξηγήσεων που έδωσα εκεί, πως η Επιτροπή Ρέτζη χρειάζεται και Χρειάζεται μάλλον να εργαστεί για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής και το έχει κάνει εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε εστιάσει την προσοχή σε αυτό το θέμα. Έχουμε επενδύσει λοιπόν σε διάφορες νομοδοτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίσματα, ε, εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και επί των ε, νομοθετικών προτάσεων που λάβαμε στις, ε, στα τέλη του Μαΐου. Τέλος, Τη Δευτέρα και την Τρίτη ε, αυτή την εβδομάδα έγινε η συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ που είναι η διάσκεψη των ε, Προέδρων των ε, Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Αυτή έλαβε χώρα στη Σόφια. Εγώ ήμουν μέρο τη αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με την κυρία Μαγκίνε, την αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, και την κυρία Τανούτα Χουμπνέρ, πρόεδρο ε, της πολύ σημαντικής Επιτροπής ΑΦΚΟ. Οπότε, τρεις εξημών συμμετείχαμε στη συζήτηση. Έγινε μια ειδική συζήτηση που εστιάστηκε στο μέλλον της πολιτικής συνοχής και πάλι εξέφρασα την θέση της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω πως αυτό ήταν πολύ χρήσιμο, διότι έτσι είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μετά από τη συνεδρίασή μας τον Νοέμβριο του 2017 ε, δουλέψαμε ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και τώρα είμαστε ιδιαίτερα ε, κινητοποιημένοι για να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές να τον αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό για να προετοιμάσουμε τη θέση της Επιτροπής Ρέτζη για τις τα διάφορα νομοθετικά ζητήματα και τις γνωμοθετήσεις μας επί άλλων ε, νομοθετικών ε, φακέλων. Αυτές είναι οι ανακοινώσει. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Φανίστερο και την κυρία Βέστφαλ για τη συμμετοχή τους, διότι έτσι ήμασταν πολύ ισχυρή ομάδα που αντιπροσωπεύσαμε την Επιτροπή μας. Αυτές ήταν λοιπόν οι ανακοινώσεις μου και τώρα συνεχίζουμε με τις κοινέ διατάξεις με τα διάφορα ταμεία το Κοινωνικό Ταμείο Πλάς, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, και τους δημοσιονομικούς κανόνες για τα ταμεία αυτά και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλειας αλλά και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και τις Θεωρήσεις CPR, έτσι το λέμε πιο σύντομα όλο αυτό. Εμείς είμαστε αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για αυτό το νομοθετικό φάκελο. υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για ψηλό επίπεδο συνεργασίας, αλλά είμαστε στην πορεία της διαπραγμάτευσης με τις άλλες επιτροπές. Και ε, σήμερα το πρωί δεδομένης της παρουσίασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Μάλλον, συγγνώμη, η Κομισιόν έχει προτείνει τέσσερις νομοθετικούς φακέλους, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτόν. Είναι ένα μακροσκελές και περίπλοκο έγγραφο, αλλά για σήμερα ζητήσαμε τον κύριο Έρικ Φον Μπρέσκο να μας το παρουσιάσει με κομψό και κατάλληλο τρόπο. Ο κύριος Φαν λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τη νομική πρόταση που υποβάλαμε πριν από δύο εβδομάδες. Είναι υψηλέ ε, οι προσδοκίες, γιατί αυτό που είπατε, το να το παρουσιάσει κανείς με κομψό τρόπο, είναι δύσκολο. Έχω προετοιμάσει μερικές διαφάνειες Συγχωρέστε με γι' αυτό. Ελπίζω να δείξετε υπομονή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, αλλά απαιτείται υπομονή. Θα διατρέξουμε μία προς μία τις ε, νομικές προτάσεις και θα σας παρουσιάσω τα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα θα εξετάσουμε τον ε, κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Πρώτα απ' όλα, ποιε είναι οι τρεις βασικές λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτή την πρόταση. Είναι ε, κάτι το σύγχρονο, η πολιτική πρέπει να είναι σύγχρονη λοιπόν, απλή, ευέλικτη. Ξέρω ότι έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για την απλούστευση, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτή τη φορά πραγματικά το εννοούμε. Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα λοιπόν, πιστέψτε με η πολιτική θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη για να ανταποκρίνεται ε, σε αναδυόμενες ανάγκες σε μια δεκαετή περίοδο ελοποίηση και τέλος πρέπει να είναι μια πολιτική για όλες τις περιφέρειες και όχι μόνο για τις πιο φτωχές. Ας ε, δούμε αρχικά το νομικό αρχιτεκτόνιμο αυτό. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων συμπεριλαμβάνει 7 ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης για να αντιποκριθούμε ε, στα παράπονα πολλών ε, δικαιούχων και αρχών που λένε ότι έχετε πολλά διαφορετικά εγχειρίδια κανόνων για τα επιμέρους ταμεία και είναι πολύ δύσκολο, μάλλον αδύνατο να τα υλοποιήσει κανείς όλα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να έχετε ένα ενιαίο εγχειρίδιο ε, για όλα τα ταμεία. Προσπαθήσαμε να το πετύχουμε. Βλέπετε εδώ ότι καλύπτονται 7 ταμεία Η κυρία Μιχαήλοβα, η πρόεδρος, ανέφερε προηγουμένω και ποια είναι τα ταμεία αυτά, αλλά θα δείτε ότι λείπει ένα. Το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη που δεν καλύπτεται από τον κανονισμό. που δεν καλύπτεται λοιπόν από την πρόταση δυστυχώ. Ε, ο κανονισμός για το ταμείο αυτό βέβαια ουσιαστικά αντιστοιχεί σε πολλές από τις διατάξεις αυτού του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Τι σημαίνει αυτό, οτιδήποτε αποφασιστεί εδώ και φυσικά και στο Συμβούλιο για αυτόν τον κανονισμό, πολλά από τα άρθρα αυτά αυτομάτως θα ισχύσουν και για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για παράδειγμα, ε, χρηματοδοτικά εργαλεία, ε, ε, εδαφική ανάπτυξη, το πρώην πρόγραμμα Leader. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν εδώ, παρότι τυπικά δεν καλύπτεται το Ταμείο. Θεωρώ όμως ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Ότι πλέον 7 ε, ταμεία καλύπτονται από έναν και μόνο κανονισμό. Τι βλέπουμε λοιπόν ε, σε αυτόν τον ε, κανονισμό. Βλέπετε εδώ στα αριστερά, πρώτα απ' όλα είναι ζητήματα ε, παράδοσης και ε, στόχων ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητα και ούτω καθεξής. Έχουμε επίσης συγχωνεύσει δύο κανονισμούς σε έναν ε, για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνεχής. Πρόκειται για διαφορετικά εργαλεία. Έχουμε συγχωνεύσει τα δύο σε ένα γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερο έτσι. Και αν δείτε τους δύο κανονισμούς, είναι ουσιαστικά το ίμιση του ισχύοντος κανονισμού σε μήκο, αν θέλετε, σε έκταση κειμένου. Προσπαθήσαμε πραγματικά λοιπόν να απλουστεύσουμε, να αποσαφηνίσουμε το κείμενο για να είναι πιο απλά τα πράγματα για όσους θα πρέπει να τα υλοποιήσουν όλα αυτά. Βλέπετε εδώ τι καλύπτεται στη μέση. Ε, θέματα, ζητήματα θεματικής συγκέντρωσης, γιατί θέλουμε οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να διοχετεύουν κάποια από τα κεφάλαια σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς στόχους πολιτικής, μετά ε, είναι θέματα αστικής ανάπτυξης και μετά για τις πλέον απόμακρες περιοχές. Έχουμε διατάξεις ε, εξόχως ε, από περιοχές, έχουμε λοιπόν ε, ιδιαίτερες διατάξεις για αυτά. Το τρίτο πακέτο θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, αφορά τη συνεργασία. Και εδώ έχουμε ουσιαστικές αλλαγές. Αν δείτε τη συνεργασία, δηλαδή τον κανονισμό Interreg, μία θεμελιώδης ε, αλλαγή που θα παρουσιάσω στη συνέχεια είναι ότι πλέον έχουμε συμπεριλάβει και τα στοιχεία εκείνα που καλύπτουν τη συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι γνωρίζετε περισσότερο αυτή την κατάσταση, θα ξέρετε ότι έχουμε διαφορετικά εργαλεία. Από πλευράς μας έχουμε μεικτή διαχείριση και το ERDF ε, το Περιφερειακό Ταμείο από τη δική μας πλευρά των συνόρων. Από την άλλη πλευρά των συνόρων έχουμε διαφορετικές ε, δομές. Αν πρόκειται για υποψήφιες χώρες έχουμε ε, για το μέσο βοήθειας προενταξιακής, αλλιώς είναι η πολιτική γυτνίασης. Πλέον θα υπάρχει ένα ενιαίο εγχειρίδιο και στα εξωτερικά σύνορα. Να μην έχουμε δύο ή τρία διαφορετικά για αυτές τις ε, περιοχές και καταρχήν ε, η υλοποίηση και διαχείριση των Ταμείου θα γίνονται με βάση τους δικούς μας κανόνες. Μεκτή διαχείριση λοιπόν, κάτι το οποίο δεν υπάρχει για τα εξωτερικά σύνορα. Και πάλι λοιπόν σημαντικό ε, δείγμα προόδου. Η πιο καινοτόμως από όλες τις προτάσεις είναι αυτό που βλέπετε το ECBM ο Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Μηχανισμό Πρόκειται για ένα νέο νομικό εργαλείο που επιτρέπει στις αρχές που βρίσκονται στα σύνορα να εφαρμόσουν το νόμο γειτονικού κράτους μέλους για την υλοποίηση αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε νομικά προσκόμματα στα σύνορα και θα θέλαμε εδώ για συγκεκριμένα διασυνοριακά έργα προκειμένου να επιταχύνουμε την υλοποίηση, οι δύο αρχές που συνεργάζονται να ε, εφαρμόσουν μόνο τις, τους κανόνες του ενός κρατούς μέλους ή του άλλου ε, για το συγκεκριμένο έργο. Και αυτό είναι ε, σημαντική καινοτομία, αλλά θα επανέλθω στη συνέχεια. Δύο λόγια τώρα για τους στόχους πολιτικής. Μίλησα για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Βλέπετε εδώ ότι θα έχουμε 5 αντί για 11 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά βέβαια αφορούν την καινοτομία, την ε, οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, συνδεσιμότητα, κοινωνική Ευρώπη και κάτι πρόσθετο εδώ, κάτι καινούριο, η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες βιώσιμη ανάπτυξη σε πόλεις, στην Ήπεθρο, στις ε, παράκτιες περιοχές. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένους ε, στόχους, ένα συγκεκριμένο στόχο που μπορούν να επιλέξουν όσοι διαχειρίζονται τα προγράμματα για να λύσουν τα ζητήματά τους. Δεν χρειάζεται λοιπόν από διαφορετικά τμήματα του κανονισμού ε, να επιλέγουν συγκεκριμένα σημεία για να καλύψουν τα ζητήματά τους. Έχουμε έναν ρητό νέο στόχο υπαριθμών 5. Δεξιά βλέπετε ότι κάθε από, κάτω από κάθε έναν ε, στόχο πολιτικής έχουμε και οριζόντιους στόχους. Πρώτον, πρέπει να βελτιώσουμε την διοικητική ικανότητα όσων διαχειρίζονται και εφαρμόζουν τα προγράμματά μας. Στον κάθε ένα από αυτούς τους στόχους, λοιπόν, ε, συμπεριλαμβάνεται και αυτή η διάσταση της οικοδόμησης δυναμικού στα κράτη-μέλη, σε περιφέρειες και σε πόλεις. Το δεύτερο οριζόντιο μέτρο είναι συνεργασία μεταξύ περιφερειών και διασυνοριακά. Γιατί βλέπουμε ότι σε πολλά από τα σημερινά προγράμματα ε, υπάρχει μια σωστρέφεια πάντα. Εμείς θέλουμε το αντίθετο. Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, ακόμα και διασυνοριακά. Και αυτό θα καταστεί δυνατό στο μέλλον υπό κάθε μία από αυτές τις πολιτικές. διατηρήσαμε αλλά εξορθολογήσαμε αυτό που λέμε τώρα εξάντε όροι για να βελτιώσουμε τις, ε, τους κανόνες ε, επενδύσεων. Έχουμε περιορίσει τον αριθμό. Πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε 35, υπερβολικός αριθμός, και τους έχουμε κατεβάσει σε 20. Με πολύ σαφέστερη ε, σύνδεση με την πολιτική. Η σημερινή εξάντε αιρεσιμότητα αφορά περισσότερο την ε, εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών που ε, κατά το μάλλον ή τον συνδέονται με τα ταμεία μας. Θεωρούμε όμως ότι αν υπάρχει όντως ένα πρόβλημα με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών, αυτό θα πρέπει να επιλύεται με διαφορετικά μέσα, διαδικασίες υποπαραβάση και το καθεξής και να επικεντρωθούμε σε, αυτές, ε, σε αυτούς τους κανόνες αρεσιμότητας, είτε είναι στρατηγική φύση, είτε όχι, για να διασφαλίσουμε την επιτυχία αυτών των ταμείων. Έχουμε λοιπόν κάπως ε, αποσαφηνίσει τη σύνδεση με την πολιτική και τέλος έχουμε περιορίσει το διοικητικό άχθος. Αυτή τη στιγμή αν ένα κράτος μέλος δεν πληρεί την εξάντα ρεσιμότητα, πρέπει να καταρτήσει ένα μακροσκελές σχέδιο δράσης που μετά το συζητάει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ γραφειοκρατία, <coughs> δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ε, κόβονται πια τα σχέδια δράσης, τα προγράμματα δράσης. Περιορίζουμε και του την εξάντα ρεσιμότητα ε, και η Επιτροπή σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου και όχι μόνο στην αρχή θα προσδιορίζει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις. Γιατί λόγω διοικητικών ή άλλων αλλαγών μπορεί κάποιο κράτος να προσφέρει καθυστέρηση. Στα δεξιά της διαφάνειας βλέπετε και άλλες ε, προϋποθέσεις ε, σαφής ε, και ισχυρή σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό σημαίνει ότι στα προγράμματα που θα υιοθετηθούν, ελπίζουμε ήδη από την αρχή, ε, το 2020, 2021 το αργότερο, θα δούμε σε ποιο βαθμό οι επενδύσεις αφορούν και, και εστιάζονται και στις ειδικές αναχώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υπάρχει ήδη ακόμα μάλλον η μακροοικονομική αιρεσιμότητα που ξέρω ότι δεν είναι πολύ δημοφιλής ε, στο Κοινοβούλιο. Το έχουμε και αυτό το μέσο εξορθολογήσει, έχει γίνει πιο ευφυές αν θέλετε. Όσοι συμμετείχαν σε προηγούμενη υπόθεση όπου μιλούσαμε για ε, αναστολή ε, της εκταμείευσης κονδυλίων για την Πορτογαλία και την Ισπανία, η διατύπωση είναι ατυχής γιατί δεν αφήνει κανένα ε, περιθώριο στην Κομισιόν να καταλήξει κατά πόσο έχει νόημα ή όχι, είναι σκόπιμο, γιατί είναι υποχρεωτική ε, ρητή η οχι ειναι σκοπιμο γιατι ειναι υποχρεωτικη ρητη διαταξη shall. Ε, πλέον υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προχωρήσει σε τέτοια αναστολή, εάν θεωρήσει ότι δεν είναι κατάλληλη η λύση. Παραμένει λοιπόν η μακροοικονομική αιρεσιμότητα, αλλά είναι λίγο πιο ε, ευφυής πλέον ε, και η διατύπωση. Διασύνδεση υπάρχει και με το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει η Επιτροπή μέχρι το 2020, αλλά και πάλι αυτό δεν αφορά μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, οριζοντίως αφορά όλο τον ενωσιακό προπολογισμό πρόταση για την τήρηση του κράτους δικαίου. Η χρηματοδότηση λοιπόν μπορεί να ανασταλεί σε αντίθετη περίπτωση. Όμως αυτό δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τη δική μας ε, πρόταση. Αφορά γενικά όλο τον ενωσιακό προπολογισμό. Σας είπα πολλά για την ε, απλούστευση. Εμείς έχουμε εντοπίσει 80 τέτοια στοιχεία απλούστευσης, αλλά δεν θα τα πω όλα τώρα εδώ. Ε, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε την εξέταση και εγχειριδίου χρήσης. Ε, ήθελα μόνο να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, και εδώ είχαμε και τη στήριξη του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις Omnibus ε, για να ε, σταματήσουμε να εργαζόμαστε με τιμολόγια και το καθεξής και κατά βάση να ασχολούμαστε με να δουλεύουμε με καταποκοπήν ποσά και το καθεξής. Ένα παράδειγμα που και πάλι θεωρώ ιδιαίτερα καινοτόμο Σήμερα πληρώνουμε, καταβάλουμε τέλη τεχνική συνδρομής σε προγράμματα ε, για την ε, συλλογή των ε, εισιτήριων λεωφορείων, των χρονοδιογραμμάτων, υπογραφή διάφορων εγγράφων. Στο μέλλον αυτό δεν θα είναι απαραίτητο. Γιατί λέμε ότι ο σκοπός της τεχνικής συνδρομής είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων. Πώς μετρούμε την υλοποίηση των προγραμμάτων με την αποστολή προς την Επιτροπή ε, ετήσεων αποζημίωσης. Για κάθε 100 ευρώ που θα ζητάτε αποζημίωση, εμείς θα σας πληρώνουμε αυτομάτως και ένα top-up, 2,5% ε, νομίζω για το ERDF, 4% για το ESF, μέχρι και 106-7 ευρώ λοιπόν, χωρίς κάποιο αποδεικτικό. Αυτομάτως λοιπόν θα επιστρέφονται ε, αυτά τα έξοδα. Δεν θα απαιτείται πλέον όλη αυτή η χαρτούρα που είχαμε προηγουμένως. Αυτό είναι μια σαφής βελτίωση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία με μικρή προσταθεμανιαξία, αξία, ε, ενώ τώρα πάμε σε μια απλουστευμένη διαδικασία χωρίς κανένα διοικητικό άκθος. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να περιορίσουμε το διοικητικό άκθος κατά 25% με αυτό το μέτρο. Δεύτερον, σήμερα μεγάλη δυσκολία ε, μας δημιουργεί ε, το κατά πόσο ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ή όχι. Και υπάρχει πάντα μια διαμάχη με τα κράτη-μέλη, ερμηνεύουμε, περαιρμηνεύουμε. Με την Πολωνία είχαμε πρόσφατα τέτοια ζητήματα, δεν θέλω να επεκταθώ, ε, αλλά υπάρχουν διάφορες δομές παράκαμψης ή μη επιστροφής του ΦΠΑ που πλέον αντικαθίστανται από έναν πολύ απλό κανόνα. Για όλες τις εργασίες που είναι κάτω των 5 εκατομμυρίων είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ χωρίς ε, ε, περαιτέρω αποδείξεις και εξηγήσει. Το 96% όλων των προγραμμάτων συνοχής είναι κάτω από το ε, όριο αυτών των 5 εκατομμυρίων. 96% έτσι. Εκεί δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τον ΦΠΑ. Είναι επιλέξιμος αυτομάτως. Για όλα τα προγράμματα επιχειρήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων, όμως δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ. Πολύ απλός ο κανόνας, ε, σαφώς και θα υπάρξει συζήτηση για το κατόφλι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλή η κατάσταση σε σχέση με σήμερα, όπου είναι πολύ δύσκολο πάντα να αποφασίσουμε. Ουσιαστικά κάθε μήνα ε, τίθεται αυτό το ζήτημα με τα κράτη-μέλη. Δεν θα έχουμε κανόνες για ε, την ε, παραγωγή εσόδων. Νομίζουμε ότι οι σημερινοί κανόνες και για τους, ε, θα έρθουν στους συντελεστές χρηματοδότησης καλύπτουν το επιπλέον διοικητικό άχθος που είναι απαραίτητο για τους διαχειριστές των προγραμμάτων να δείξουν και να αποδείξουν κατά πόσο υπάρχει υπερβολική χρηματοδότηση ή όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες πια, ε, διαγράφονται. Αντίστοιχα και ε, η έγκριση των, μεγάλων προγραμμάτων από την Επιτροπή. Έτσι κι αλλιώς ε, ήταν λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Θα έχουμε μια νέα κατηγορία προγραμμάτων, προγράμματα στρατηγικής σημασίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι μεγάλα σε μέγεθος, μπορεί να είναι και μικρά, αλλά πρέπει να είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Εδώ, σαφώς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα επιλέξουν, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, να υποβάλουν εκθέσεις και να τα δημοσιοποιούν. Όμως, και πάλι μπορεί να είναι από οποιοδήποτε κλάδο, γιατί σήμερα κυρίως αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται στο περιβάλλον και στις μεταφορές, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε και άλλους κλάδους και να εντοπίσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά προγράμματα. Αλλά δεν θα εγκρίνονται από την Επιτροπή πια, θα είναι η ε, διαχειριστική αρχή ε, και η Επιτροπή Παρακολούθησης. Μετά κάτι που είναι πραγματικά ρεξικέλευθο και μας πήρε πολύ καιρό να πείσουμε τους συναδέλφους εντός της Επιτροπής, ε, δεν υπάρχει πια η διαδικασία ε, διορισμού. Ε, πολλές φορές καθυστερούσαμε γιατί καθυστερούσε όλη η διαδικασία διορισμού από την εθνική αρχή. Στο μέλλον δεν θα υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία ή πρώτερος έλεγχος. Ουσιαστικά ε, θα εγκρίνουμε τις ε, αρχές του προγράμματος όσα έχουν και αν ε, αλλάξει κάτι, τότε η ελεγκτική αρχή θα είναι αυτή που θα πρέπει να κάνει έλεγχο, όπως οφείλει, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία διορισμού. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και πάλι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα άρδιν είναι ότι θα κάνουμε ένα βήμα πίσω ε, για τα προγράμματα με χαμηλά ποσοστά σφάλματος, για τα τρέχοντα προγράμματα. Για παράδειγμα, αν ένα πρόγραμμα το 2021, που είναι ένα πρόγραμμα που διαδέχεται ένα άλλο που υπάρχει ήδη το 19-20, και έχει αποδείξει το 19 και 20 ότι έχει χαμηλό ε, ποσοστό σφάλματος ή παρατυπιών, ε, μπορεί να μας ενημερώσει το πρόγραμμα ότι σε ό,τι αφορά την επαλήθευση ε, από πλευρά διαχείριση θα εφαρμόζει μόνο εθνικού κανόνε. Και αυτό είναι σημαντική αλλαγή. Μέχρι τώρα είχαμε δύο σύνολα κανόνων. Ενωσιακοί, ενωσιακοί κανόνε διαχείριση, έλεγχη κτλ. και τους εθνικούς κανόνες για την εθνική χρηματοδότηση. Όπως ξέρετε, στην περίπτωσή μας ε, έχουμε και τα δύο γιατί υπάρχει συγχρηματοδότηση. Πλέον λοιπόν τα κράτη-μέλη μπορούν να ελέγχουν ε, τις δαπάνες βάσει των εθνικών κανόνων μόνο και Επιπροσθέτω σε ό,τι αφορά τους λογιστικούς ελέγχου, δεν χρειάζεται να κάνουν ελέγχου συστήματος, μόνο μερικές ε, επιχειρήσεις κάθε χρόνο για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί το σύστημα. Είναι σημαντική αυτή η βελτίωση. Δεν κοιτάζουμε τα κρατημέλη, κοιτάζουμε τα προγράμματα. Οπότε, ενδεχομένως, να ισχύσει αυτή η διάταξη για όλα τα προγράμματα στην Ένωση και όχι μόνο για μερικέ ε, χώρε. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο λειτουργεί το πρόγραμμα ή όχι. Και υπάρχει κάτι ακόμα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά θα επανέλθω. Είπα προηγουμένως ότι βασικός στόχος είναι η ευελιξία. Και θέλω εδώ να επισημάνω δύο ζητήματα. Βλέπετε πάνω-πάνω. Αυτή τη στιγμή για κάθε τροποποίηση του προγράμματο πρέπει να υποβάλει αίτηση τροποποίηση προγράμματο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κράτου να το κοιτάξει η Κομισιόν, να ξεκινήσει μια διαδικασία τροποποίηση. Αυτό παίρνει πολύ καιρό και είναι ιδιαίτερα επαχθή διαδικασία. Στο μέλλον, αν έχουμε ίσονο σημασία τροποποιήσεις, δηλαδή μόνο 5% των κονδυλίων ε, πηγαίνουν από τη μία προτεραιότητα στην άλλη, τότε η διαχειριστική αρχή μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να ζητήσει έγκριση από την Κομισιόν. Απλώς μας ενημερώνει. Έχουμε μετατοπίσει τα κονδύλια από εδώ προς τα εκεί. Ε, υπάρχει αυτή η αλλαγή, αλλά δεν απαιτείται έγκριση ή κάποια επιπλέον διαδικασία. Δεύτερον, ε, η πρότασή μας να έχουμε ενδιάμεση αναθεώρηση το 2025. Τι σημαίνει αυτό. Οι διαχειριστές των προγραμμάτων μπορούν τώρα να πραγματίσουν τα πρώτα πέντε έτη, αλλά όχι το 2026 και 2027. Παγώνουν αυτά τα έτη στα προγράμματα. Και σκοπός είναι να επανέλθουμε το 2024-2025 και να συζητήσουμε αν έχουμε νέες ανάγκες. Για παράδειγμα, μεταναστευτικό και εκεί θα υπάρχει, δυνατότητα να μετατοπίσουμε τη χρηματοδότηση από τη μία προτεραιότητα στην άλλη. Και υπάρχει ε, και μία νέα ε, δυνατότητα μεταβίβασης ορισμένου μεριδίου ε, της χρηματοδότησης σε άλλα μέσα. Τώρα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιδόσεις και τους ε, ελέγχους αξιολογήσης. Θα περιοριστώ μόνο να πω ότι καταρχάς θα μειωθεί το αποθεματικό επιδόσεων, το οποίο θεωρούμε πως ε, δεν είναι τόσο αναγκαίο, μια που θα αντικατασταθεί από την διάμεση αναθεώρηση το 2024 και 2025. Φεύγει λοιπόν αυτό από τον κανονισμό και επίσης φεύγουν οι ε, ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση μέχρι το τέλος Ιουνίου περίπου δημοσιεύονται αυτές οι εκθέσεις που καλύπτουν το προηγούμενο έτος. Τώρα δηλαδή θα λάβουμε ε, τις εκθέσεις για το 2017. Τώρα αυτό θα συμβεί σε 300 και παραπάνω προγράμματα συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και μετά σας στέλνουμε μία έκθεση περιληπτική περίπου τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο του 2018 σχετικά με την ε, κατάσταση υλοποίησης που όμως καλύπτει το περασμένο έτος. Στο μέλλον θεωρούμε πως θα πρέπει να περάσουμε σε ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων έτσι ώστε η πολιτική συνεχίζει να περάσει στον 21ο αιώνα. Και επίσης ε, να γίνεται ουσιαστική συζήτηση στις συναντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση με τα κράτη-μέλη, όπου θα γίνονται ε, ερωτήσεις επί της ουσίας. Δεν θα υπάρχει όμως αυτή η ανταλλαγή αρχείων PDF που είναι έτσι κι αλλιώς ε, παροχημένη. Επίσης, αυτό που φεύγει είναι η υποχρέωση διεξαγωγής εκ των ε, προτέρων αξιολόγησης Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κομμάτι όπου θα αναφέρονται τα διδάγματα που αντλήσαμε και τα συμπεράσματα που ε, βγάλαμε για το τι θα γίνει σχετικά με το μέλλον, αλλά το σημαντικό είναι ε, ότι ενισχύεται ο ρόλος των ε, επιτροπών ελέγχου, αυξάνεται η διαφάνεια και ε, σχετικά με τον ε, κώδικα διοντολογίας, ίσως θυμάστε πως ήταν κάτι καινούργιο για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε διάφορες έρευνες σύμφωνα με τις οποίες απεδείχθη πολύ χρήσιμος ο κώδικας διοντολογίας. Τον στήριξε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως ε, είχε έρθει με καθυστέρηση για συγκεκριμένα προγράμματα και χρειάστηκε χρόνος μέχρι να γίνει ο συντονισμός, να επιλεγεί η κατάλληλη διατύπωση κτλ. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα διατηρήσουμε τον ε, υφιστάμενο κώδικα διοντολογίας, δεν θα αλλάξουμε τον κανονισμό και τα προγράμματα θα μπορούν να αρχίσουν να καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση όπως έχει σήμερα. Αυτό λοιπόν θα μείνει, δεν αλλάζει και αρχίζει να υπολογίζεται ήδη από τώρα. Δεν έχει γίνει λοιπόν καμιά τροποποίηση. Υπάρχει μια μετακύληση αν θέλετε στην επόμενη περίοδο, εφόσον δεν υπάρχει ε, ανάγκη για αλλαγές. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκαν οι απαιτήσει ε, για τη διαφάνεια και για ε, την προβολή των προγραμμάτων. Ήδη αναφέρθηκα σε αυτά τα νέα project που είναι στρατηγικής σημασίας όπου τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να διεξάγουν διάφορες ε, δραστηριότητες και εκδηλώσεις ε, προβολής, έτσι ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση του κοινού, να αυξηθεί η διαφάνεια. Όλα σε ένα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την κατάσταση. Νομίζω πως πήγαμε ε, ένα βήμα παραπέρα, ακριβώς διότι τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά και δε αυτή την εποχή είναι δύσκολο να πείσουμε τους πολίτες για την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ε, να περάσουμε στην ε, αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Εδώ έχει γίνει μια γενικότερη ευθυγράμμιση. Δεν θα αναφερθώ τώρα στι εκ των προτέρων αιρεσιμότητε. Ε, θα πω μόνο ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή και είναι ιδιαίτερα καινοτόμο αυτή η αλλαγή ε, η δυνατότητα να συνδυάζουν τα χρηματοδοτικά μέσα με επιχορηγήσει μέσω ενό νέου μηχανισμού. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν υπάρχει ένας ε, χρηματοδοτικός μηχανισμός, και υπάρχουν δύο ε, project, υπάρχουν και δύο διαφορετικές αρχές που ε, συνδέουν τους δικαιούχους με ε, τα χρήματα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο δίνει μια επιχορήγηση στον δικαιούχο ή η τράπεζα χορηγεί ένα δάνειο. Στο μέλλον αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν, δηλαδή θα μπορεί να χορηγείται δάνειο και επιχορήγηση και ελπίζουμε αυτό να οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις, διότι αυτή τη στιγμή αυτά γίνονται ξεχωριστά. Θα υπάρχει λοιπόν μία υπηρεσία, μία αρχή που θα κάνει και τα δύο και θεωρούμε ότι αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα ακριβώς διότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσε να αποβεί πάρα πολύ χρήσιμο να ενωθούν ε, οι δύο αυτές λειτουργίες σε μία. Θα απλουστεύσει επίσης τις ε, πληρωμές, όμως δεν θα πω σε λεπτομέρειες, γιατί αυτές ε, διέπονται από άλλους απλουστευμένους κανόνες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Επίσης, γνωρίζετε ότι τώρα υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων και ταμείων. Εμείς πάμε ακόμα παραπέρα γιατί όπως γνωρίζετε το ΕΕΦΣΙ θα αντικατασταθεί από ένα άλλο επενδυτικό ταμείο όπου τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε αυτό μέχρι 5% των ε, πιστώσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η απλούστευση εδώ έχει να κάνει με το ότι η συνεισφορά αυτή θα συνεχίσει μεν να αφορά στόχους συνοχής, αλλά θα εφαρμόζονται μόνο οι κανόνες του Invest EU. Θα υπάρχει δηλαδή ένα νέο σύστημα κανόνων. Διότι προς το παρόν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα και πολλά κράτη-μέλη δυσκολεύονται στο να εφαρμόσουν τα συστήματα αυτά. Θα γίνεται λοιπόν ε, μεταφορά, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που θα αναφέρονται στα προγράμματα, όμως τα κονδύλια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ε, κανόνες του InvestEU. Τώρα, στο, στη διαφάνεια υπάρχει και ένα παράδειγμα ε, που μπορείτε να δείτε. Το πρώτο παράδειγμα, το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει στην Επιτροπή, ε, υπάρχει το πρόβλημα των ε, επικαλύψεων και έχει συζητηθεί το θέμα του καλύτερου συντονισμού. Εδώ έχουμε νομίζω καταλήξει σε, σε μια πάρα πολύ καλή πρόταση την ε, ευρωπαϊκή αριστεία στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό. Εάν υπάρχει ένα πρόγραμμα αριστείας, ένα έργο το οποίο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του ε, προγράμματος ορίζοντα, αλλά δεν έχει επαρκή κονδύλια, τότε η αρχή διαχείρισης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία για να στηρίξει ε, τον ε, δικαιούχο του προγράμματος αυτού. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι ότι αυτό στην ουσία δεν λειτουργεί και γιατί, διότι οι κανόνες είναι πολύπλοκοι. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει και με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι ότι αυτά τα έργα θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία χωρίς ε, περαιτέρω απαιτήσει. Δεν θα υπάρχουν και δεν θα εφαρμόζονται κανόνες ε, για τις κρατικές ενισχύσεις στην περίπτωση αυτή. Θα υπάρχει δηλαδή η ίδια μεταχείριση ε, όπως και στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα θα υπάγονταν στον ορίζοντα. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι δυνατόν διότι τα διαρθρωτικά ε, ταμεία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά δεν θεωρείται κράτος και γι' αυτό το πρόγραμμα ορίζοντας ε, δεν θεωρείται ε, πως συμμορφώνεται με τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις. Συμφωνήσαμε όμως ότι στο μέλλον αυτά τα project θα χρηματοδοτούνται αυτόματα από τα διευθυντικά ταμεία και θα ε, διέπονται από τους ίδιους κανόνες που διέπουν και τους κανόνες της κρατικές ενισχύσεις. Τώρα, θα απαντήσουμε τα χαρά σε ερωτήσεις για αυτά. Αλλά να περάσω στο βασικό μας θέμα, το χρήμα. Και εδώ είναι δύσκολο να περιοριστώ σε λίγα λόγια. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω λέγοντας ότι γνωρίζουμε ότι έχει περικοπεί κατά 10% ο προπολογισμό της πολιτικής συνοχής. Δυστυχώς, όμως ε, αυτό δεν είναι απόφαση δική μου, οπότε δεν μπορώ να το σχολιάσω. Σίγουρα όμως με το νέο μικρότερο προπολογισμό είχαμε τρεις στόχους. Πρώτον, να ε, επικεντρωθούμε ε, στους ε, φτωχότερους, τα κράτη-μέλη με τις περισσότερες δυσκολίες. Έπειτα, η πολιτική μας στις πιο αναπτυγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει νόημα και αντίκτυπο. Δηλαδή για κάποιες περιφέρειες της Δανίας, του Βελγίου, των κατοχωρών, σε αυτές τις περιοχές που είναι ήδη αναπτυγμένες αρκεί να γίνουν κάποιες απλούστερες προωθητικές ενέργειες. Και τρίτον, θέλαμε να περιορίσουμε τις ε, απώλειες από την αλλαγή ανάμεσα στην ε, υφιστάμενη και τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, όπως ξέρετε, να περάσει και στο Συμβούλιο, διότι χρειάζεται ομοφωνία για να εγκριθεί. Τι έχουμε κάνει λοιπόν. Στην ουσία διατηρήσαμε την υφιστάμενη μέθοδο πιστώσεων, τη μέθοδο του Βερολίνου όπως λέγεται. Όπως βλέπετε το ΑΕΠ είναι ο πιο σημαντικός δείκτης. Βλέπουμε ότι πάνω από το 80% των κονδυλίων πιστώνεται σύμφωνα με το ΑΕΠ και οι αλλαγές ε, που θα γίνουν είναι πολύ μικρές. Ε, παρομοίως με την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή ε, απασχόληση, επίπεδο εκπαίδευσης κτλ. Ούτε εδώ αλλάζει κάτι. Εδώ έχουμε εισαγάγει δύο νέα στοιχεία. Πρώτον, για τη μετανάστευση. Και αυτό γιατί στο μέλλον η μακροπρόθεσμη ένταξη των μεταναστών θα είναι ένας από τους στόχους της πολιτικής συνοχής και θέλαμε να φανεί. Και δεύτερον, επειδή θέλαμε να ε, δώσουμε έμφαση σε επενδύσεις για το περιβάλλον, έχουμε εισαγάγει και το περιβάλλον. Βλέπουμε όμως ότι το συνολικό βάρος των πρόσθετων πιστώσεων είναι μηδαμινό. Μετά προσαρμόσαμε κάπως και τις τρεις κατηγορίες περιφερειών. Παραμένουν τρεις. Εδώ βλέπετε τον χάρτη που έχουμε σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι φυσικά υπάρχουν, και υπάρχουν παραμένουν οι αναπτυγμένες περιοχές, οι μεταβατικές και οι λιγότερο αναπτυγμένες, όμως έχει γίνει μία αλλαγή. Έχουμε περάσει από το... 75% ε, στο 100% των ε, περιφερειών. Και γιατί. Διότι, σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει, όλες οι περιφέρειες που βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ανεβαίνουν σιγά-σιγά, βελτιώνονται. Οι πιο φτωχές στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχουν τάσεις βελτίωσης και βρίσκονται από το 75% στο 85%. Νομίζω η μόνη ε, περίπτωση που έχει σημειωθεί απώλεια 8% είναι στις περιφέρειες που βρίσκονται στο 90% των ε, του ποσοστού ανάπτυξης και θα ήταν πιστεύω κρίμα να μην μπορούμε να ε, δώσουμε σημαντική στήριξη και να ανεβάσουμε τα ανώτατα όρια στο 100%. Έτσι θα εποφεληθούν ορισμένες περιφέρειες διατηρώντας το, την κατηγορία της ε, μεταβατικής περιφέρειας από περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, για παράδειγμα στις χώρες της Βαλτικής, Τσεχία, Πολωνία. Οι περιφέρειες αυτές ε, παίρνουν πορτοκαλί χρώμα, το οποίο καταδεικνύει η βελτίωση. Βλέπετε ότι στην Ελλάδα οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ορατές, η χώρα έχει γίνει σχεδόν όλη πορτοκαλή, η Νότια Ιταλία ολόκληρη και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στο Ταμείο Συνοχής, ισχύει η επιλεξιμότητα που υπάρχει σήμερα. Βλέπουμε τις χώρες με μόβ χρώμα που είναι επιλέξιμες για το Ταμείο Συνοχής. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν κάτι. Τέλος, σίγουρα στη διαφάνεια δεν βλέπετε τα νούμερα γιατί είναι πάρα πολύ μικρά. Εδώ βλέπουμε τις πιστώσεις ανακράτος μέλος και θα δείτε ίσως τις αλλαγές ανάμεσα στις δύο περιόδους προγραμματισμού. Βλέπουμε λοιπόν και τις ε, αλλαγές ε, στη, στα νούμερα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι, ορισμένες χώρες που έχουν ε, χάσει μέχρι και το 25% των πιστώσεών τους. Θεωρώ όμως πως αυτό πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διότι Μία χώρα σαν την Ισπανία, για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό έχασε το 45% των ε, πιστώσεων. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, 25 δισεκατομμύρια περίπου. Έχουμε λοιπόν ε, δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, ε, το μείον 24%, το οποίο θα περιορίσουμε τις αλλαγές ανάμεσα στις δύο περιόδους προγραμματισμού, έτσι ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες. Όμως αυτό φυσικά μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω και τέλος θα δείτε και τα νούμερα στην ε, πρότασή μας στη σελίδα 22 αν δεν κάνω λάθος θα δείτε και την ανάλυση ε, ανακράτος Τώρα, γιατί δημοσιεύσαμε αυτά τα στοιχεία. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχει διαφάνεια και σίγουρα αυτό το θέλει και το Κοινοβούλιο και θέλει επίσης να έρθει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο πριν τις επόμενες ευρωεκλογές. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ε, την πρωτοβουλία να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, κάνουμε το πρώτο βήμα, ε, παρουσιάζουμε ευθύ εξ αρχή την κατάσταση και ελπίζουμε αυτό να μας εξοικονομήσει κάποιο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε με λεπτομέρειες στο Συμβούλιο τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα συμβεί στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με διαφάνεια ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, έχω λίγα ακόμα πράγματα να σας πω. Πρώτον, ποσοστά συγχρηματοδότησης. Μπορείτε εδώ να δείτε τα στοιχεία στις οθόνες σας. Ε, η πρότασή μας είναι να μειωθούν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Γιατί? Πρώτον, για να αυξηθεί η ανάληψη ευθύνης και η οποία φυσικά ε, όταν έχεις επενδύσει δικά σου χρήματα αυξάνεται αυτόματα και έπειτα ε, επειδή τα ποσοστά συγχρηματοδότησης είναι ακόμα πολύ ψηλά ως ε, αντίκτυπος της ε, κρίσης. Στην Ελλάδα για παράδειγμα υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά, 90-100% ε, συγχρηματοδότηση μετά το 2021 θα αλλάξει αυτή η προσέγγιση και επιθυμούμε να επιστρέψουμε σε πιο φυσιολογικά ποσοστά, τα οποία θα αυξήσουν το γενικότερο αντίκτυπο της συνεισφοράς μας. Ελπίζουμε να έρθει σε μια ισορροπία κατάσταση γιατί θα μειωθούν, θα μειωθούν τα ποσοστά, θα αυξηθούν τα ποσοστά της κρατικής χρηματοδότησης. Αυτό θα γίνει με την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας. Για παράδειγμα, ΦΠΑ αν θέλουμε να αποζημιώνουμε, επιστρέφουμε το ΦΠΑ χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό κρατών μελών, ε, θα πρέπει να είμαστε λιγότερο ευέλικτοι από τις άλλες διατάξεις. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι περισσότερη κρατική χρηματοδότηση, αλλά δίνουμε και μεγαλύτερη ευελιξία σε ορισμένα θέματα που αφορούν την υλοποίηση, όπως για παράδειγμα αιρεσιμότητα, ε, ΦΠΑ. Κλείνουμε δηλαδή εντό αγωγικών τα μάτια για ορισμένες περιπτώσεις. Και τέλος, προτείνουμε να επιστρέψουμε στον ΙΣΙΝ 2 διότι στην τρέχουσα περίοδο έχουμε παρατηρήσει ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων στην παρούσα περίοδο γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και ε, αυτό οφείλεται εν μέρη στον κανόνα νησιν 3. Δεν θέλουμε να πάμε στον νησιν 3 από την αρχή. Θέλουμε αυτό να γίνει σταδιακά σε ένα πρώτο στάδιο να πούμε ότι για τον πρώτο χρόνο ε, θα έχουμε μόνο 60% ε, πιστώσεις, μετά θα αλλάζει το ποσοστό, θα ανεβαίνει κατά 10 κτλ. Θα παρέχεται λοιπόν περισσότερη ευελιξία στα κρατημέλη και στα προγράμματα αυτά έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινούν πολύ γρήγορα την υλοποίησή τους, δεν θα υπάρχει ε, αρχή εξουσιοδότησης, όμως και εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιούνται τα προγράμματα χωρίς να περιμένουμε χρόνια, δύο-τρία χρόνια μέχρι να αρχίσει το στάδιο της υλοποίησης. Δίνουμε λοιπόν μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση. Ταυτόχρονα ζητάμε όμως και να λάβουν τα κράτη-μέλη αυτή την ευελιξία στα σοβαρά. Θα σταματήσω όμως εδώ, να ζητήσω συγγνώμη για την ε, μεγάλη παρουσίαση και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Σας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε και Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και οι πληροφορίες που μας δώσατε. Θέλω να σας θέσω μια ερώτηση. Ε, θα κάνετε άλλη παρουσίαση για το RDF ε, ε και για τη συνοχή και για τα... Ναι, α, μάλιστα. Έχουμε δύο ώρες και 20 λεπτά για συζήτηση, εφόσον δεν έχετε άλλη παρουσίαση. Και έχουμε, και έχουμε τρεις ακόμα παρουσιάσεις και τρεις ακόμα συζητήσεις, οπότε θα βάλω όρια για τις ερωτήσεις. Γιατί... Ε... 1,5 λεπτό ο καθένας. και να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες παρουσιάσεις. Λοιπόν, αρχίζουμε με τους συντονιστές, διότι όλοι έχουμε ορίσει εισηγητές. Ε, και ο κύριος Βάνιστερ πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. σημερινή συνεδρίαση είναι περισσότερο ενημερωτική, όπως είπαμε, όπως βλέπω. Οπότε πιθανό πως ε, δεν πρέπει να έχουμε ήδη συμπεράσματα. Είναι σωστό αυτό που είπατε. Ε, δεν, ε, όλοι οι εισηγητές είναι γνωστοί. είναι επικεφαλής, έχουν αρχίσει να δουλεύουν, είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Είναι σημαντικό να έχουμε την ε, ταχύτητα που χρειάζεται ε, και είναι καλό να έχουμε αυτή την ε, ενημέρωση από την Κομισιόν να προχωρήσουμε στις πολιτικές συζητήσεις και επαφές με τους εισηγητές που γίνονται ταυτόχρονα Ήδη δηλαδή μπαίνουμε με πέφτουμε με τα μούτρα στη δουλειά για να ασχοληθούμε με εκείνα τα τμήματα της πρότασης που μπορεί να αποφασιστούν φέτος σε αυτή την Επιτροπή. Μπορεί να έχουμε δηλαδή ήδη την πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να έχουμε δέσμευση στην Επιτροπή, αλλά ίσως το 90% των πραγμάτων να μπορούν να γίνουν και μάλιστα μπορεί και σε fast track. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι από τους ηγητές μας πριν από το καλοκαίρι κιόλα να έχουν ε, καταθέσει το έγγραφό τους για μετάφραση και να κάνουμε τις προφορικές μας τροποποίησεις στις πρώτες εβδομάδες Σεπτεμβρίου. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί αν ακούσουμε προσεκτικά, πολλά έχουν ήδη γίνει. Ήδη έχουν αναπτυχθεί πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Αν αρχίσουμε να ασχολούμαστε με κάθε λεπτομέρεια θα χάσουμε χρόνο. Έχω μία ερώτηση μόνο. Έχουμε δει στοιχεία για τα κράτη-μέλη και νούμερα. Θα ήθελα να ξέρω πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα κριτήρια και τα νούμερα. Πόσο έχω δει, τα νούμερα των κρατών μελών χρησιμοποιούνται. Το θέμα είναι, υπήρξε μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τα αποτελέσματα, ειδικά αυτοί που που μειώνονται τα ποσά τους. Έχει γίνει καμιά διαπραγμάτευση ή είναι κάπου μεταξύ. Δεν καταλαβαίνω. Μήπως ο κ. Βανπρέσκα μπορεί να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που κρατήσατε και το χρόνο σας πάνω κάτω. Κυρία Μπρέσο, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Βέστφαλ που μου το επιτρέπετε γιατί η κυρία Μπρέσο πρέπει να φύγει. Ευχαριστώ. Έχω μια παράλληλη συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΚΟ και είμαι σκιώδης για μια, για μια εισήγηση εκεί. Ε, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση που μας κάνατε. Έχω μια ερώτηση. Επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω καταρχάς ε, αυτές τις διαφάνειες που μας παρουσιάσατε γιατί θα μας χρησιμεύσουν για να μπορέσουμε να ε, συνοψίσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα στοιχεία. Δεύτερον, ε, θελοντική συμβολή στο InvestEU είναι μία συμβολή των κρατών, ή, όχι των περιφερειών, ή μπορούσαν να είναι και οι περιφέρειες, όπου δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Τρίτον, βλέποντας τα στοιχεία πολλών χωρών, αυτό που προκύπτει είναι ότι οι πρωτεύουσε εστιάζουν όλο και περισσότερο, μάλλον συγκεντρώνουν όλο ένα και περισσότερο πλούτο. Ακόμα και στις χώρες όπου το ε, μεγαλύτερο κομμάτι των περιφερειών είναι κάτω από το 50% ξαφνικά φτάνουν στο 130-140% στις ε, πρωτεύουσες. Αν το κοιτάξει κανείς δηλαδή, για παράδειγμα η Μπρατισλάβα έχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρώπης, πιο ψηλά και από τη Στοκχόλμη. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Οι πιο απομακρυσμένες περιφέρειες ε, όλο ένα και περισσότερο ζημιώνονται από τις, περιφέρει... από τις πρωτεύουσες γιατί πάντοτε ξεπερνούν το μέσο όρο. Κάποιες φορές αυτό είναι και ανεξάρτητο από το ευρωπαϊκό κονδύλια, ε, αλλά από την άλλη έχουμε σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, μεγάλη πιθανότητα να, υπάρχουν, να υπάρχει και συγκέντρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. το έχετε λάβει αυτό υπόψη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Βέστεφαλ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση έχω μόνο σχετικά με την κρατική διάσταση. Πριν από δύο χρόνια ψηφίσαμε όντως όλα αυτά που είπατε και τώρα συνειδητοποιούμε ότι με τις νέες προτάσεις το 85% των κονδυλίων πηγαίνουν σε, στις πλουσιότερες περιοχές, σε προγράμματα για το περιβάλλον κτλ. και δεν μένουν πολλά για τις υπόλοιπες. Αυτό νομίζω πως είναι αντιπαραγωγικό ε, ιδιαίτερα μάλιστα σε σχέση με αυτό που ψηφίσαμε πριν από δύο ε, χρόνια, γιατί όχι, που ψηφίσαμε ότι όχι μόνο οι πόλει, αλλά και οι ε, ύπεθρος θα πρέπει να δέχονται ενισχύσει. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω κάποια μεγαλύτερη ευελιξία. Γνωρίζω πως, πως υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων, όμως κάποτε πρέπει να γίνει η αρχή. Και η αρχή θα πρέπει να είναι όντως ε, το ότι θα πρέπει να δούμε την αστική διάσταση λίγο διαφορετικά, ακριβώς ε, διότι υπάρχουν και οι περιαστικές περιοχές τις οποίες δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Τόμασιτς. κυρία Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα περισσότερα που ακούσαμε σήμερα και διαρωτώ με για τις ε, γιατί κάποιες χώρες αυτό το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνα είναι η εθνική συμβολή. Γιατί σύμφωνα με τη νέα πρόταση το ποσοστό της χρηματοδότησης είναι 30% για τις χώρες και το 70% της χρηματοδότησης προέρχεται από την Επιτροπή. Πώς στάσαμε σε αυτά τα ποσοστά. Ευχαριστώ, Very much. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως είναι μια πολύ καλή προσέγγιση να έχουμε περισσότερη ευελιξία και τελικά και περισσότερη εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Όλες αυτές οι ανταλλαγές ε, δείχνουν πως πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα σχόλια μας για την επόμενη περίοδο λοιπόν θα πρέπει να είναι περισσότερο σχετικά με το τι θα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Ευφυής εξειδίκευση. Έχουμε πρώτα τις προτεραιότητες, τους παλιούς φακέλους, μετά τις νέες προτεραιότητες Και έπειτα έχουμε και τα, κονδύλια για τις ε, ειστερούσες περιοχές, γιατί μέχρι στιγμή σε αυτή την προοπτική στα κράτη-μέλη είχαμε ένα λειτουργικό πρόγραμμα σε περιφερειακό επίπεδο. Και έπειτα ένα θέμα που αφορά το εργαλείο 5+, τι σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή αν μια χώρα εξαντλήσει τελείως τα κονδύλια που έχει για μια προτεραιότητα, τότε αυτό το εργολείο επιτρέπει την άμεση χρήση των υπόλοιπων δύο. Στην Κροατία, ας πούμε, χρησιμοποιούμε την προτεραιότητα 3 για τις μικρομεσαίες και κοντεύει αυτό το κονδύλι να εξαντληθεί. Αν λοιπόν δύο χρόνια δεν έχουν εξαντληθεί, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους επιπλέον πόρους αμέσως για τις μικρομεσαίες. Αυτή η ευελιξία αυτό σημαίνει είναι μόνο για έκτακτες περιστάσεις. Και έπειτα για την συγχρηματοδότηση το 70% είναι πολύ χαμηλό για τις λιγότερο αναπτυγμένε ε, χώρες, η συνάδελφος το είπε ήδη, και η ε, αντικατάσταση της επιλεξιμότητας ε, ΦΠΑ δεν νομίζω ότι είναι σωστή, γιατί είναι 70% των επιλέξιμων δαπανών και σε πολλές περιπτώσεις είναι μόνο 30 ή 40% του επίπεδου του project. Χρειάζεται κάτι παραπάνω λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσίαση. Όσο μπαίνουμε στις λεπτομέρειες βέβαια, τόσο περισσότερα ερωτήματα ανακύπτουν. Εφόσον δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα περιοριστώ μόνο σε ένα ζήτημα, το θέμα των ε, συνεργειών. Λέτε στην πρότασή σας ότι οι ε, προτάσεις ε, προγραμμάτων που έχουν λάβει τη σφραγίδα ε, της αριστείας από το ορίζον δεν χρειάζεται να περάσουν άλλη μία διαδικασία επιλογής από το ERDF. Αυτό μήπως είναι όμως απλώς όνειρα θερινές νυχτός, γιατί και για τις κρατικές ενισχύσεις τι γίνεται. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι κανόνες εθνικών επιδοτήσεων δεν ισχύουν για αυτό το πλαίσιο. Ε, τι γίνεται με τον περιπολογισμό που θα παίρνει διαθέσιμος. Σε κράτη-μέλη με λιγότερα κονδύλια κάποια στιγμή φαντάζομαι για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ουσιαστικά δεν θα υπάρχει προϋπολογισμός. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εφόσον έχει λάβει σφραγίδα αριστεία από την Κομισιόν, αυτομάτω παίρνει χρηματοδότηση από το ERDF, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό τη Κομισιόν εδώ. Ένα δεύτερο, για, για την αναθεώρηση επιδόσεων. Έχει αντικατασταθεί πλέον από το 5 2. Τι κάνει όμω η Κομισιόν όταν το κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τις ειδικέ αναχώρας συστάσεις στα προγράμματα από την αρχή και μετά από πέντε χρόνια ε, έρχεται αντιμέτωπο με νέες ειδικέ αναχώρας συστάσεις ε, και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη και έχει την πολιτική βούληση να πει όχι αναστέλουμε την ε, χρηματοδότηση για τα επόμενα δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Όλμπριχτ. Uh, ένα γενικό σχόλιο. Γιατί είμαι και εισηγητή ε, για το ΠΔΠ. Και ένα ερώτημα. Το σχόλιο. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ε, για τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε. Γιατί το νέο κεφάλαιο δεν ε, αντανακλά το προηγούμενο κεφάλαιο. Από κάτω λένε παραδοσιακή πολιτική και μιλούν για τρία ταμεία. Όταν συγκρίνουμε το 75% και τις λιγότερες, ε, ε, λιγότερα αναπτυγμένες είναι μόνο δύο ταμεία. Γιατί μιλάμε λοιπόν δύο, τρία ταμεία. Πείτε μας. Από πολιτική άποψη, βέβαια, όταν κάποιο θέλει να πετύχει έναν στόχο, ε, ακολουθεί μια μέθοδο και χρησιμοποιεί δείκτε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αντικειμενικούς δείκτες και αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης, όχι το αντίστροφο. Να ρωτήσω λοιπόν, γιατί το Ταμείο Συνοχής έχει υποστεί μείωση 46%. Προσπαθώ να το κατανοήσω. Καταλαβαίνω ότι περισσότερο θα πάνε στο ERDF στις ε, περιοχές μετάβασης, περιφέρειες μετάβασης. Αλλά γιατί να πάρει λιγότερη χρηματοδότηση το Ταμείο Συνοχής. Και τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Invest in You» ε, Γιατί υπάρχει πρόταση προαιρετικά, εθελοντικά, να πάρουμε χρήματα από εκεί και να τα πάμε στα λεγόμενα Windows που δεν θα υπάρχει τίποτα για τη συνοχή αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε τα χρήματα θα φύγουν από τη συνοχή, θα πάνε στο «Invest in You» και τι γίνεται με τις κρατικές ενισχύσεις. Γιατί σε ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας δεν υπάρχει ε, κρατική ενίσχυση, ενώ... Τέλος πάντων, δεν το έχω καταλάβει, ρώτησα και τον κύριο Κατάινεν, πείτε μου εσείς. Ευχαριστώ κύριο Σφίκο. Ευχαριστώ, <clears throat> Πρόεδρε. Και εγώ στηρίζω την ε, την παρουσίαση αυτή και θεωρώ πως αυτή, αυτός ο κανονισμός ε, πρέπει να μελετηθεί εις βάθος και να συζητηθεί ε, βέβαια σύντομα αλλά αποτελεσματικά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Είδαμε ότι εστιαστήκαμε περισσότερο στα οικονομικά θέματα αλλά θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να δούμε και ε, το ζήτημα της πιστοποίησης κάνουμε κάποιες αρχικές παρατηρήσεις για κάποια σημεία τα οποία είναι θετικά, όπως η μεγαλύτερη συγκέντρωση των στόχων, όπως η ενίσχυση του ρόλου των πόλεων και των περιφερειών ή η διοικητική απλοποίηση. Θέλω ωστόσο να θέσω σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη συνδέεται σε, με μια αξιολόγηση που δηλώθηκε ρητά όσον αφορά το πώς θα δοθούν ε, οι χρηματοδοτήσεις. Αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί με τις χώρες και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης επίσης έχουν ήδη συμφωνηθεί. Έπειτα, μήπως θα αντιμετωπίσουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, αν η αύξηση της συγχρηματοδότησης ε, της εθνικής ε, μπει μέσα στο σύμφωνο σταθερότητας, τότε θα πρέπει να δούμε πως τα κράτη δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες ε, που οδήγησαν στο μπλοκάρισμα της χρήσης αυτών των ε, πόρων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν επίσης την τροποποίηση των χρόνων ελέγχου. Μήπως υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν αποσαφηνήσεις όσον αφορά το θέμα κάθε ταμείου, κάθε προγράμματος, κάθε δίκαιση που είναι αρμόδια να υπάρχει μια αρχή διαχείρισης, μια πιστοποίηση και μια ελέγχου γιατί υπήρξαν σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια για να δούμε μήπως η πρόταση απλοποίησης στην οποία αναφερθήκατε είναι ε, ε, αποτελεσματική όχι, γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Άνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Φανπρέσκα για αυτήν την λεπτομερέστατη παρουσίαση της ε, πρότασης της Επιτροπής. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τις ερωτήσεις της δικής μου πολιτικής ομάδας. Ε, καταρχάς, για τους ε, πράσινους, ε, το Ταμείο είναι κυρίως για την ενίσχυση, για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτή την ενοποιημένη προσέγγιση. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χωρίσει αυτά τα δύο από τον γενικό κανονισμό. Ενώ μάλιστα μας λέτε πώς πρέπει να γίνει αποδοτικότερη χρήση των ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων. Μετά, ε, η... στην πολιτική συνοχή στηρίζουμε την ε, κοινωνική διάσταση και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το ποσοστό που θα ε, μεταφερθεί από το ε, ESF. Έπειτα, μας είπατε για πλούστευση και μας αναφέρατε ορισμένα στοιχεία, ε, όμως αναρωτιέμαι Πού πήγαν ε, τα υπόλοιπα. Μας είπατε ότι απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες, όμως εγώ βλέπω ότι κάποια στοιχεία εξαφανίστηκαν τελείως. Έχουν περάσει σε μεταγενέστερη φάση υλοποίηση. Υπάρχει ε, κάποια προσθετικότητα εξαρτώντα από προϋποθέσεις. Εμένα μου φαίνεται πως ε, δεν πρόκειται εδώ για πλούστευση, αλλά για ριζική αλλαγή, για αναρδιάρθρωση, η οποία έχει πολιτική ε, προέλευση και φυσικά και πολιτικές επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω πώς εσείς μπορείτε να διασφαλίσετε την ισότητα, την ε, απαγόρευση των διακρίσεων στην υλοποίηση προγραμμάτων και γιατί έχετε, αλλά, έχετε κάνει τις αλλαγές που έχετε κάνει έπειτα. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως αποστασιοποιείται από την ανάληψη ευθυνών στα μεγάλα έργα. Γιατί όμως, ε, ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής και ποιος θα είναι ο μελλοντικό της ε, ρόλος σε αυτά τα μεγάλα έργα. Ο έλεγχος ε, λέτε πως ε, δεν είναι τόσο ε, αναγκαίος που μετακυλίεται το βάρος του, αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι τα χαμηλά ποσοστά χρηματοδότησης, ε, οι μειώσεις που θα γίνουν, οι αυξανόμενες απαιτήσεις προς τα κράτη-μέλη και αυξανόμενες απαιτήσεις επίσης ε, προς τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Εδώ θα υπάρξουν προβλήματα, διότι είναι μεν υπάρχουν ε, οι πιο εύπορες περιφέρειες, αλλά υπάρχουν και οι φτωχότερες οι οποίες θα συναντήσουν τεράστιες δυσκολίες. Ευχαριστώ. Να επενθυμίσω ότι υπάρχει πολύ στενό χρονοδιάγραμμα σας παρακαλώ λοιπόν να τηρείτε το χρονικό σας όριο. Κύριε Ντεμάτο. Ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω κατευθείαν τις ερωτήσεις μου. Παραμένει η σύνδεση ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δυστυχώ η θέση δεν έχει αλλάξει, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα σε σχέση με τον προγραμματισμό τη ε, μακροαιρεσιμότητα. Έχει αλλάξει η δυνατότητα να ανασταλούν οι πληρωμέ εάν ανασταλούν οι δεσμεύσει στι περιφέρειες των χωρών που δεν σέβονται του συγκεκριμένου προγραμματισμού αναχώρα, το εξάμεινο δηλαδή. Έπειτα, από τη μια πλευρά λέμε ότι πρέπει να είμαστε φυσικά η Ευρώπη της υποδοχής, όμως η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει πάλι ακόμα μια φορά να ε, τιμωρηθεί με επενδύσεις για την άμυνα και την ασφάλεια. Γιατί η δική της αναλογία είναι τελείως διαφορετική και ο στόχος είναι διαφορετικός και θα πρέπει να είναι τελείως ξεχωριστή. Ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ξέρουμε πως ε, στην ουσία η Επιτροπή Απασχόλησης είναι αρμόδια επί της ουσίας, αλλά θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι διαθετικές ε, μεταρρυθμίσεις δεν έχουν σχέση με την πολιτική συνοχή κανονικά υπό το φως του προγράμματος 23 εκατομμυρίων ευρώ που συνεχίζει να προτείνει η Κομισιόν. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται αυτός ο σύνδεσμος. Είμαστε και εμείς κατά της μείωσης ε, της συγχρηματοδότησης γιατί παραμένουν οι δεσμεύσεις του, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και άρα ε, εκτός και αν δεν θέλουμε να παρέμβουμε με τα μία τα διαρθωτικά για τον που, δεν... Ε, ε, υπολογίζονται ως έλλειμμα. Ε, περιμένω λοιπόν οι τροπολογίες που όλοι μας θα υποβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση θα εγκριθούν και θα μπουν στη συμβιβαστική. Γιατί τώρα το Ταμείο για την Ανάπτυξη Υποέθρου έχει βγει από το ρυθμιστικό πλαίσιο και για τα χρηματοδοτικά μέσα. Είναι σημαντικά και θα είναι όλο και πιο σημαντικά. Άρα λοιπόν η επιλογή τους είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να γίνονται και κερδοσκοπικά. Τα equity, τα trust fund, τα άλλα είδη ομολόγων, το έχουμε ήδη πει επανειλημμένα, ότι θα ήταν χρήσιμο και λογικό να υπάρξουν εγγυήσεις και ε, ε με συγκεκριμένα επιτόκια, ακόμα και αν είναι ε, με μακρά τα διαστήματα αποπληρωμής. Επίσης, να διευκολυθούν οι τύποι ε, peer-to-peer, ε, crowdfunding και social lending. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην θέλει κανείς άλλο το λόγο. Θα δώσουμε μόνο το λόγο στον συνεισηγητή, κύριο Νοβάκοφ. Κύριε Κρέλε δεν είναι εδώ, οπότε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω αρχικά τους διερμηνείς ε, για τη δουλειά που κάνουν εδώ και για τον κύριο Βανμπρέσκο για την παρουσίασή του. Έχω μια σειρά ερωτήματα. Για μένα δεν ήταν σαφές ε, κατά πόσο οι τιμέ είναι σταθερές ή οι τιμές από την αρχή της προγραμματική περίοδου για να κάνουμε σύγκριση. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί ε, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υιοθέτηση της πρότασης, Έχοντα κατά νου ότι μένει ακόμα ένας χρόνος πάνω κάτω για να ολοκληρωθεί. Και την περασμένη φορά μα πήρε τρία χρόνια σχεδόν. Θα μπορούσατε να μας ε, ενημερώσετε και για το Ταμείο των Μικρών Προγραμμάτων. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Ε, πώς ε, θα το διαχειριστείτε και τι είδους αποτελέσματα περιμένετε. Τέλος, θεωρείτε ότι η σύμβαση του Ταμείου Συνοχής στην διευκόλυνση της συνέντασης στην Ευρώπη θα πρέπει σε αυτό το βαθμό να αφήσει το Ταμείο Συνοχής με 30 δισεκατομμύρια. Θεωρείτε ότι αυτό το ποσό φτάνει για τη στήριξη όλων των επιλέξιμων δικαιούχων του Ταμείου Συνοχής για 7 χρόνια και για πολύ σημαντικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αυτά ήταν τα ερωτήματα των Ευρωβουλευτών για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Το λόγο έχει ο κύριος Φων Βρέσκο. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ερωτήσεις. Είναι και καιρός πιστεύω να δώσουμε και τις κατάλληλες απαντήσεις. Θα τις ε, πάρω από την αρχή και θα πω καταρχάς πως συμφωνώ με τον κύριο Βανίστελ Ρόι. Αυτό Άλλωστε προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα θετικά στοιχεία και μια σταθερότητα. Και επίσης ε, στα καλά αυτά στοιχεία ανήκουν και αυτά που πήραμε από τον κανονισμό Omnibus. Ε, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε ε, κρατήσει, κώδικας διοντολογίας για παράδειγμα και τα υπόλοιπα που, που αναφέρθηκαν. Θα ήθελα όμως να τονίσω την απλούστευση Έγινε δημόσια διαβούλευση πριν την κατάρτιση της πρότασής μας και φάνηκε ένας γενικότερος, μια γενικότερη ανησυχία για το θέμα της ανάγκης απλούστευσης των ε, περίπλοκων ε, κανόνων. Καταλήξαμε λοιπόν στο ότι πρέπει να παρέμβουμε εκεί που χρειάζεται και να ε, μην ε, είμαστε υπερβολικά παρεμβατικοί. Να κάνουμε λοιπόν ένα βήμα πίσω και να δούμε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Τώρα θεωρώ πως θα έπρεπε να απαντήσω τώρα και στην ερώτηση του κυρίου Νόβακοφ, ε, αν έχει δηλαδή νόημα να ξαναδούμε τα κομμάτια του κανονισμού που θα παραμείνουν και να δούμε πώς χρειάζονται αλλαγές. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, και ελπίζω να συμφωνήσει και το Συμβούλιο, ε, τα οποία νομίζω πως ε, θεωρούμε όλοι σωστά, νομίζω πως ε, πρέπει να βασιστούμε στα, σε αυτά που, που έχουμε κοινά και να προχωρήσουμε, διότι όσο καθυστερούμε τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τα προγράμματα να υλοποιηθούν, διότι δεν θα υπάρχει καμία ασφάλεια δικαίου. Ε, αυτό είναι προς απάντηση στον κύριο Νόβακο. Χρειάζεται συνεργασία το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να ε, υλοποιηθεί η πρόταση. Τώρα, κύριε Βανίστελ προς το παρόν δεν έχει γίνει ε, κάποια συζήτηση για το ποιου δείκτες θα χρησιμοποιήσουμε κτλ. Αυτό που είδαμε είναι πως υπήρξαν διάφορες ενστάσεις από τα κράτη-μέλη, διάφορα παράπονα διότι έλεγαν πως δεν είχαν ε, όλες τις πληροφορίες που χρειάζονταν, πως δεν ήταν ικανοποιημένα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, Έχουμε εισαγάγει αρκετούς δείκτες για το κλίμα, για τη μετανάστευση και αυτό πιστεύω αντανακλά και αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την πολιτική μας, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τις ελλείψεις στους τομείς αυτούς και να βοηθήσουμε τις περιφέρειες εκείνες και τα κράτη-μέλη εκείνα που χρειάζονται στήριξη, που πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους ε, ε, τομείς αυτούς. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί νέοι δείκτες που ε, περιγράφουν αυτές τις ανάγκες και νομίζω πως ε, δημιουργήσαμε και αυτά τα δίχτυα ασφαλείας, ότι δηλαδή κανείς δεν μπορεί να έχει απώλειες πάνω από 4%. Βέβαια, στην ε, τρέχουσα περίοδο το ποσοστό είναι μείον 45%. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν δραστική μείωση του ε, ποσοστού ασφαλείας αλλά το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι να περιοριστούν οι απώλειες. Ε, διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο πολιτικά να ε, περάσει μια τέτοια πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνουν όλα αυτά έτσι ώστε να περάσουμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Κύριε Μπρέσο, ρωτήσατε πώς λειτουργεί το EU Invest. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή όπου οι περιφέρειες και τα κρατημέλη πρέπει να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν την επιμερισμένη διαχείριση για τα χρηματοδοτικά μέσα ή να περάσουν από το InvestEU επειδή το θεωρούν ε, καλύτερο. Και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα από την αρχή να ε, καταδείξουν τι ποσά θέλουν να μεταφερθούν στο InvestEU έτσι ώστε να επιτευχθούν ποιοι στόχοι πολιτικής. Αυτό αναφέρθηκε ε, νωρίτερα. Οι λόγοι είναι ε, για λόγους ε, συμμόρφωσης Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω πως αυτό το θέμα ίσως αφορά περισσότερο ε, χώρες όπου αντιμετωπίζουν θέματα διοικητικά. Επίσης υπάρχει και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ορισμένων κρατών μελών που ε, διαφέρει στα κράτη-μέλη. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό κακό, κανείς δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα. Τώρα, οι διαφορές ανάμεσα στις ε, πρωτεύουσες, στα μεγάλα κέντρα και ε, στην Ήπεθρο έχουν να κάνουν με το ότι θέλουμε να δώσουμε περισσότερη ευελιξία στη μεταφορά κονδυλίων. Αυτή τη στιγμή μόνο το 3% μπορεί να μεταφερθεί, αλλά στο μέλλον το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί, θα πάει στο 15% από τη μία, προς τη μία κατεύθυνση και ε, θα είναι απεριόριστη, απεριόριστο το ποσοστό μεταφοράς ε, προς την άλλη κατεύθυνση. Φυσικά υπάρχουν και άλλες νομικές διατάξεις που θα διέπουν αυτές τις μεταφορές, όμως αυτή τη στιγμή δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Ε, το σχόλιο τώρα της κυρίας Βέστφαλ για την αστική ανάπτυξη ε, να ε, επιστρέψω τώρα στην αρχική μου παρουσίαση, να σας παραπέμψω σε αυτή και να πω ότι υπάρχουν ελαφρώς μεγαλύτερες πιστώσεις για την αστική ανάπτυξη. Προσπαθούμε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και αυτό είναι κάτι που ε, αφορά κυρίως τα αστικά κέντρα. Μετά, αρκετοί από εσά έκαναν την ίδια ερώτηση για το από, από πού προέρχονται τα στοιχεία μας. Ε, λοιπόν, καταρχάς υπάρχει ε, η αρχή της ανταπόδοσης. Ε, δεν θα υπάρχουν πλέον διατάξεις που θα αφορούν ε, τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Αυτό που θα γίνει είναι πως ε, κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέφεται ο ΦΠΑ, θα χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο ε, κάποια έργα διότι δεν υπάρχουν διατάξεις για την δημιουργία ε, εσόδων. Όμως, όπως είπαμε και πριν, θα περάσουμε σε ποσοστά συγχρηματοδότησης ε, που υπήρχαν ε, στην εποχή πριν την κρίση. Το ανώτατο ποσοστό ήταν 75% τότε και ο ΦΠΑ δεν ήταν κατά ανάγκη επιλέξιμος. Θέλουμε λοιπόν να επιστρέψουμε στην περίοδο πριν την κρίση και νομίζω πως το 2021 θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να το κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, νομίζω πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ε, μόνο προς τα πάνω μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ίσως το Συμβούλιο συμφωνήσει γρήγορα, αλλά μάλλον θα συμφωνήσει για το ότι το βάρος θα πρέπει να περάσει από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μάλεβιτς, για την ε, τοπική ανάπτυξη δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές, τα πράγματα παραμένουν όσα έχουν. Σε ό,τι αφορά την ευφυή e εξειδίκευση, να σας πω ότι καλύπτεται από τον ε, στόχο πολιτικής 1. Είναι πολύ βασική αυτή η αλλαγή. Ότι υπό την ε, στρατηγική της εφιούς εξειδίκευσης στον στόχο 1, τα κράτη-μέλη και οι διαχειριστές προγραμμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα, ε, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να ενισχύουν διάφορες δεξιότητες ε, για δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Διότι ακριβώς χρειάζεται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να υπάρξει ανάπτυξη. Και αυτό πρέπει να γίνει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και θεωρούμε πως ε, θα ήταν πολύ χρήσιμο να ε, υπάρχει χρηματοδότηση από ένα ενιαίο μέσο. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την FEE εξειδίκευση και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων γιατί είναι μία από τις δαπάνες ε, τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί. Θα περάσω τώρα στις ερωτήσεις του κυρίου Όλμπριχτ για τον αριθμό των ταμείων. Αναφέρομαι στα ταμεία που υπάρχουν στην πολιτική συνοχή, στο, στο περιφερειακό ταμείο. Όμως, τα διάφορα συστατικά στοιχεία της πολιτικής ε, συνοχής έχουν και διαφορετικές ε, μεθόδους επιστώσεων. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τέσσερις διαφορετικές τέτοιες ε, μεθόδους με διαφορετικούς ε, υπολογισμούς ε, κατανομής πόρων. Τώρα, γιατί μειώθηκε το Ταμείο Συνοχής. Δεν είχαμε τιμωρητική προσέγγιση. Το Ταμείο Συνοχής αυξήθηκε τεχνητά για τα κράτη-μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004 ή και αργότερα. Και γιατί αυξήθηκε τεχνητά κατά το 1 τρίτο, διότι χρειάστηκαν ε, βασικές ε, επενδύσεις σε θέματα υποδομής περιβαλλοντικά και περιβαλλοντικά. από το 2004 μέχρι το 2023 θα έχουμε μια περίοδο περίπου 20 ετών κατά την οποία έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις σε ε, σημαντικές υποδομές. Σίγουρα πρέπει να συνεχίσουν οι επενδύσεις στις υποδομές, όμως θεωρούμε ότι στο μέλλον ε, οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν κυρίως την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την ενεργειακή απόδοση και άλλα τέτοια, άλλους τέτοιους τομείς. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει μέσω του Ταμείου Συνοχής. Δεν θα υπάρχει λοιπόν τεχνητή αύξηση του Ταμείου Συνοχής, θα υπάρχει μία ανακατανομή των πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη και στο κοινωνικό ταμείο. Δεν θα έχει λοιπόν κανέναν απολύτως αντίκτυπο στην γενικότερη χρήση των κονδυλίων. Ήδη απάντησα στην ερώτηση του πώς μπορεί το InvestEU να το κάνει αυτό. Τώρα η σύνδεση με την εθνική συγχρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν μηχανισμό σταθερότητας. Δεν ξέρω αν το Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί ε, σύντομα με αυτό. Θα σας αναφέρω όμως εν συντομία ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ω εξή. Αν υπάρχει κάποιο κράτος μέλος που ε, έχει οικονομικές, δημοσιονομικέ δυσκολίες, το πρώτο που θα γίνει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει πρώτα την, εθνική πολιτική συνοχής. Θεωρούμε πως αυτό θα στείλει ένα σαφές μήνυμα. Έπειτα θα στηριχθούν εθνικές επενδύσεις σε τομείς επιλέξιμους ε, για την πολιτική συνοχής. Έτσι λοιπόν διασφαλίζουμε ότι αν υπάρχουν δυσκολίες από πλευράς καρτών μελών, ε, αυτές ε, θα καλυφθούν με τη στήριξή μας. και αυτό ίσως εξηγεί τα υψηλά ποσοστά εθνικής ε, χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ε, μεγάλα ελλείμματα. Μετά, ε, με ρωτήσατε γιατί βγήκε το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθυνου. Δεν έχω κάποια απάντηση. Δυστυχώς, το μόνο που θα μπορούσα να σας πω ίσως είναι ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα αλλάξει ριζικά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε στάδιο μεταρρύθμισης, θα υπάρχει μια προσέγγιση βάση στόχων που θα διέπει όλον τον κανονισμό και σύμφωνα με αυτό, εάν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για ε, το Ταμείο Ανάπτυξη τη Υπαίθρου εκτό πλαισίου κοινή γεωργική πολιτική, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο η μεταρρύθμιση αυτή να είναι, να είναι ουσιαστική και να, είναι, και να έχει συνοχή σε όλου του επιμέρου τομεί. Γι' αυτό λοιπόν ε, βγήκε το ταμείο αυτό. Θεωρούμε πως ε, πρέπει λόγω της συνοχής να εξεταστεί σε άλλο πλαίσιο. Νομίζω δεν έχουν μείνει πολλές ερωτήσεις ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε από το 375 δισεκατομμύρια τα 100 να ε, πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στην πρότασή μας λοιπόν έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αυξάνεται να σας πω κιόλας. Επίσης η κυρία Βάνα αν δεν κάνω λάθος, ρώτησε γιατί δεν αναφερόμαστε στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν θέλαμε να επαναλάβουμε στον κανονισμό τα αυτονόητα. Φυσικά και πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της μεταχείρισης και στις ε, κρατικές συμβάσεις. Βέβαια, αν δούμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας έργων θα δείτε ότι υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό. Ε, αναφέρεται για παράδειγμα ότι όταν θα επιλέγονται προγράμματα θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η ε, αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Αντί δηλαδή να υπάρχει κάποιο άρθρο στην αρχή για τις γενικές αρχές, ε, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στον τομέα της επιλογής έργων και νομίζουμε πως αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό από μια γενικότερη διάταξη. Τέλος. Η κυρία Νταμάτο μας ρώτησε για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Φυσικά και παραμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ έχει προβλέψει κάποια ασφαλιστική δικλίδα έτσι ώστε να μην μπορεί να αναστείλει τη χρηματοδότηση. Δεν θα υπάρχει βέβαια ολική εξαφάνιση αυτής. Όταν ας πούμε εισαγάγεις νέες προϋποθέσεις πρέπει να είσαι συνεπής σε όλους τους τομείς. Αυτό βέβαια είναι κάτι που έχει συζητηθεί και σε επίπεδο επιτρόπων, όπου και λήφθη η απόφαση. Και τέλος, ε, κύριε Νόβακοφ, τα στοιχεία που σας παρουσίασα αφορούν την περίοδο από την αρχή της κρίσης. Θέλουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό στους διάφορους επιμέρους τομείς του κανονισμού και να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς το συντομότερο. Ιδιαίτερα οι πιο σημαντικοί, αυτοί για παράδειγμα που αφορούν τη διαχείριση προγραμμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Και στην επόμενη παρουσίαση για το Interreg θα απαντήσω στην τελευταία σας ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις λεπτομερείς σας απαντήσεις. Νομίζω πως έτσι κλείσαμε το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί ήταν η παρουσίαση για το CPR. Τώρα συνεχίζουμε με την παρουσίαση για τις κοινέ διατάξεις, με τις ειδικέ διατάξεις μάλλον. Σταματάει η Πρόεδρος. Ναι. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής. Αυτό είναι το επόμενο. Να θυμίσω το χρόνο, το χρόνο μας. Μπορείτε να είστε λίγο πιο σύντομος. Για να είμαστε και εμείς σύντομες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω δύο λεπτά, άντε τρία. Just, uh, uh, so, uh, one thing. I already explained the policy objectives. Ε, ήδη εξήγησα τους στόχους ε, της πολιτικής. Ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ, Πρώτα θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε ένα ζήτημα που είναι νέο. Και είναι το γεγονός ότι έχουμε προτείνει στον κανονισμό δείκτες, κοινούς δείκτες για αποτελέσματα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, διότι αν δούμε τα περισσότερα προγράμματα αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιούν ειδικού δείκτες για τα προγράμματα που δεν μπορούν να, ομοδοποιηθούν. δεν μπορούν να Δεν μπορούν να μας πούν ε, ακριβώς ε, τι συμβαίνει, ακόμα και σε επίπεδο της, της χώρας και είναι πολύ δύσκολο εκ τούτου να αποδείξουμε την προστιθέμενη αξία και είναι πολύ δύσκολο να τα βάλουμε σε μια βάση δεδομένων. Γι' αυτό στο μέλλον θέλουμε να έχουμε ε, κοινούς δείκτες όσο γίνεται περισσότερο. για να είναι πιο εύκολο να κάνουμε αναφορές. Κάτι ακόμα, το ανέφερα και πριν. Θέλουμε να εστιάσουμε τουλάχιστον τμήμα των χρημάτων σε ευρωπαϊκές προτεραιότητες και να εξασφαλίσουμε κρίσιμη μάζα. Έχουμε ένα, μια αναπέτηση για θεματική συγκέντρωση. Αυτό όμως που θέλουμε τώρα είναι να έχουμε περισσότερη ευελιξία για τα κρατημέλη, δηλαδή δεν θα ελέγξουμε το σεβασμό της συγκέντρωσης σε περιφερειακό επίπεδο, θα το ελέγξουμε μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και πώς το κράτος μέλος και πώς οι διάφορες ε, ε, περιφέρειες επιτυγχάνουν το στόχο είναι δική τους υπόθεση. Δεν θα το εξετάσουμε εδώ, οπότε έχουμε πάλι ευελιξία έχουμε τρεις ομάδες κατορμελών. Αυτές που είναι φτωχές κάτω από το 75% του μέσου όρου της Ευρώπης, τις ενδιάμεσες 75 με 100% και αυτές που είναι πάνω από το 100%. Και ανάλογα με το που βρίσκεσαι έχεις ψηλότερο ή χαμηλότερο χαμηλότερη απέτηση ε, συγκέντρωσης για την καινοτομία και το χαμηλό, α, χαμηλή χρήση άνθρακα. υπάρχει δηλαδή διαλλαγή, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Έχουμε και μια αρνητική λίστα πραγμάτων που δεν θα βρούμε. Και εδώ βλέπουμε μια σειρά από στοιχεία. Σαφήνεια, νομική βεβαιότητα, τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί και τι όχι. Έπειτα, το θέμα της αστικής ανάπτυξης. Έχουμε να ενισχύσουμε τις δράσεις για την αστική ανάπτυξη. Βλέπετε εδώ τα σημεία που έχουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε μια νέα πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των πόλεων, για τη δημιουργία δυνατοτήτων, καινοτόμε δράσεις, γνώση, επικοινωνία, να τα συνδυάσουμε όλα αυτά σε μια πρωτοβουλία και αυτό που πιστεύω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι να απομακρυνθούμε από την τρέχουσα πρακτική που έχει δημιουργήσει πολλές δυσκολίες γιατί σε πολλά κράτη-μέλη τα, οι πόλεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα ταμεία, τα κονδύλια, συγγνώμη. Στο μέλλον λοιπόν να επιτρέπουμε στις πόλεις είτε να προετοιμάσουν τη στρατηγική ε, ανάπτυξη στις πόλεις ή να επιλέξουν τα project, αλλά να αφήσουν τη διαχείριση σε εκείνους που μπορούν να διαχειριστούν, που είναι τα αρμόδια όργανα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η επιλογή των project και η στρατηγική ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν έχουν λόγο οι πόλεις, αλλά δεν χρειάζεται να γίνουν και διαχειριστές. Γιατί αυτό έχει δημιουργήσει δυσκολίες και καθυστερήσεις. Γιατί απλώς δεν μπορούν να είναι manager. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις πιο απομακρυνμένες περιοχές. Έχουμε διατηρήσει την ειδική χορήγηση την ειδική μάλλον κατανομή επιτρέπει να στηριχτούν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να στηριχτούν από αλλού. Τα λειτουργικά κόστη είναι ένα παράδειγμα, επενδύσεις στα αεροδρόμια είναι ένα άλλο παράδειγμα και αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως ήσασταν σύντομος. Έχουμε διορισμένο εισηγητή, τον κύριο Κοτσολίνο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι παρόν. Πώς να προχωρήσουν τώρα οι συντονιστές πρώτα. Κύριο Βανίστερο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρίμα που ο εισηγητής δεν είναι εδώ για αυτό το σημείο. Να, το λέω γιατί δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Ε, αυτό που έχω να ρωτήσω αφορά την ευελιξία, γιατί ένα κράτος μέλος δεν χρειάζεται να προτείνει αυτή την περιφερειακή επιχειρησιακή, τα επιχειρησιακά του μάλλον προγράμματα πριν να συμφωνηθούν. Θυμάμαι σε ορισμένε χώρε όταν τις επισκεφθήκαμε, διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν, ας πούμε στη Ρουμανία, γινόταν χαμός κάποιες φορές και αυτό είναι μεγάλο φόρτο, μεγάλος φόρτος εάν αυτό οδηγεί σε κεντρική διαχείριση. Μάλλον αυτό οδηγεί σε, σε, κεντρική διαχείριση γιατί έχουμε τον, κωδικό, τον κώδικα διοντολογίας και λέει ότι αν ένα έχει περισσότερη εξουσία σημαίνει πως, δεν, πως γίνεται επανεθνικοποίηση. Ποια είναι τα μέσα εξασφάλισης, οι ρήτρες ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη συνεργασία στα κράτη-μέλη και ποια είναι η θέση τώρα στις αρχές της συμφωνίας εταιρικής σχέσης γιατί τότε μπορεί να έχεις ακόμα αρκετή επιρροή ακριβώς επειδή τα κράτη-μέλη προσπαθούν να συνδυάσουν, να προσεγγίσουν τις, τις, ε, τις, τη στάση τους κάποια στιγμή θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτά. Μπορείτε αυτό λίγο να το φωτίσετε. Ακούγονται καλά όλα αυτά, αλλά να μην απογοητευτούμε στο, στο τέλος. Είναι κοινέ οι αρμοδιότητες, κοινή διαχείριση. Κυρία Βέστφαλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να στήσω συγγνώμη από τον ε, κύριο Κοζολίνα. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να προσθέσω δύο λόγια σε αυτά που ακούσαμε. Από τη μία, χαιρόμαστε πάρα πολύ βέβαια για αυτά που ακούσαμε, ότι πράγματι δηλαδή όλες οι περιφέρειες ε, θα λαμβάνονται υπόψη στο μέλλον, ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα αφορούν όλους. Από την άλλη βέβαια βλέπουμε ότι ε, γίνονται περικοπές Περικοπές μάλιστα σε όλους τους τομείς, επώδυνες περικοπές μέχρι 10% και στις πλουσιότερες περιφέρειες ε, αυτό είναι επώδυνο διότι θα ε, πληγούν ορισμένα έργα, θα έχουμε προβλήματα. Και ρώτησα πιο πριν τι γίνεται με την αστική ανάπτυξη 85% στην ε, πιο ευφυή, πιο πράσινη Ευρώπη, αυτό θα έχει πολλές επιπτώσεις. Ε, δεν θα μείνουν και πολλά για την αστική ανάπτυξη. Όμως αυτό που με ενδιαφέρει με την ε, ιδιότητα της εισηγήτριας πριν από κάποια χρόνια είναι το περιεχόμενο Σε τι συνιστάται δηλαδή αυτή η νέα αστική ανάπτυξη, ποια είναι τα ωφέλη της. Και ε, το ότι βγήκε από τον ε, γενικό κανονισμό ε, το ταμείο, όπως ακούσαμε και πριν, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Χρειάζεται προσοχή. Ήπεθρος και οι πόλεις ε, που είχαν τόσες διαφορές και, προσπαθήσαμε με τόσο κόπο να ενώσουμε να μην κινδυνεύσουν πάλι ε, και να μην έχουν προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των έργων μας. Σας ευχαριστώ. κυρία Τόμας Ετσιλίπη κύριε κυρία Βαν Μιλτενμπουργκ. Θα θέλατε το λόγο. Και εγώ έχω ένα ερώτημα. Ε, για την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, γιατί κάπου θα υπάρχουν τα αριθμητικά στοιχεία, φαντάζομαι, στο κείμενο, αλλά δεν τα βρήκα. Ποιο είναι ο προτινόμενο προπολογισμό ε, για το σύνολο τη πρωτοβουλία αυτή, πώ ε, θα γίνει η κατανομή για κάθε μία από τι τρει ενότητε, οικοδόμηση δυναμικού, καινοτόμε πράξει, έχοντα κατά νου και το σημερινό πρόγραμμα. Και τρίτη, αυτή ενότητα για την γνώση και επικοινωνία. Ουσιαστικά ποιο είναι το διακύβημα λοιπόν για τις πόλεις, ιδίως για τις αστικές ε, ε, καινοτόμες ενέργειες που θα πρέπει να παραταθούν και μετά το 2020 κατά τη Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κυρία Μιχίλς. Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου, κυρία Μίχελς. Τώρα ακούγομαι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πολύ σύντομη, διότι ήδη έχουμε μιλήσει πάρα πολύ καιρό για ένα σημείο της ημερησίας διάταξης, δεν υπάρχει λόγος να μακρηγορούμε άλλο. Βλέπουμε εδώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι λαμβάνει χώρα μία απλούστευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη τη απλουστεύει κάποιες εσωτερικές τη διαδικασίες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχεδόν το ίδιο με αυτό που ρώτησε ο κύριο Φανίστελ Ρόι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θεωρεί ότι με μια ενίσχυση της κεντρικής διαχείρισης θα ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ το βλέπω μάλιστα ακριβώς αντίθετα. Έχω μιλήσει με την Επιτροπή των Περιφερειών και να σας πω μάλιστα ότι έχουν και εκείνη την ίδια άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βάνα δεν είναι εδώ. Ο κύριος Ροπέ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μία σειρά παρατηρήσεις. Είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα σωστό συμβιβασμό για να μην χρειάζεται να αλλάξουμε εκ των υστέρων τα προγράμματα. ενα δύο πράγματα με αποσχολούν κατά βάση. Πρώτον, η απλούστευση. Είναι ένα δημοφιλές ε, θέμα, το οποίο βρίσκουμε σε όλα τα προγράμματα. Έχουμε παρατηρήσει μια τάση. Μετά από την λήψη επιμέρους ε, αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απλούστευση, τα κράτη-μέλη ε, μπαίνουν στη διαδικασία εισαγωγής επιπρόσθετων ε, δικλείδων ασφαλείας και έτσι το πρόγραμμα γίνεται όλο ένα και πιο σύνθετο και γραφειοκρατικό. Εσεί σε τι είδου διασφαλίσει μπορείτε να δώσετε από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να μην εισάγονται πρόσθετε διαδικασίε και προποθέσει από τα κρατημέλη στη συνέχεια. Δεύτερον, η χρήση των ε, κονδυλίων στο κράτος μέλο. Ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστια ανισομέρεια μεταξύ κρατών μελών, αλλά και στο, στο ίδιο το κράτος μέλος Στη Λιθουανία, για παράδειγμα, αν δείτε την περιφέρεια της πρωτεύουσα και την υπόλοιπη χώρα, ε, είναι σχεδόν τριπλάσια, ε, ε, τριπλάσια τα μεγέθη του ΑΕΠ στην πρωτεύουσα. προτίθεστε στο μέλλον να αξιοποιήσετε τα ταμεία όχι σε εθνικό επίπεδο, αλλά με βάση τις πιο πλούσιες και πιο φτωχές περιφέρειες. Γιατί διαφορετικά, αν επενδύουμε τεράστια ποσά σε πλούσιες περιφέρειες, η συνολική απόδοση των κρατών μελών μπορεί να βελτιώνεται, αλλά τα εσωτερικά προβλήματα της κάθε χώρας θα παραμείνουν στις υπόλοιπες περιφέρειες. Μετά, πήρατε μια απόφαση να υπάρξει περικοπή της χρηματοδότησης για τις ε, μεταβατικές χώρες και να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με έναν τρόπο κάπως σταδιακά και όχι ε, μια και έξω, ούτως ώστε τουλάχιστον η συγχρηματοδότηση αυτή να αυξηθεί ε, σταδιακά σε ορισμένα χρόνια. Ιδάλλως, όταν φτάνει η χώρα στην μεταβατική αυτή περίοδο, βλέπουμε ότι ξαφνικά σταματούν οι επενδύσεις και έτσι σταματούν και τα προγράμματα και τελικά ε, αυτό δεν βοηθάει τη διαδικασία. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Κύριε δεμάτο. 50% ε, των δημοσίων επενδύσεων ε, πηγαίνει σε αυτά ε, τα project. Είπαμε ήδη ότι η στρατηγική της εφιούς εξειδίκευσης αποτελεί συνεπές πλαίσιο και προσθέτει αξία. Όμως, από μια μελέτη που έχει γίνει ακριβώς από την Κομισιόν, φαίνεται πως αυτό γίνεται στις πιο αναπτυχμένες περιφέρειες. Η Επιτροπή, λοιπόν, έχει αναρωτηθεί πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική και για τις περιφέρειες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. Σημεριζόμαστε την πρόταση της ε, Κομισιόν ε, όσον αφορά τις επενδύσεις για την αστική ανάπτυξη. Προσέχουμε ιδιαίτερα αυτή τη νέα ε, πρωτοβουλία και θέλουμε να μας πείτε με ποιο τρόπο θα υπάρξει συνδυασμός ανάμεσα σε αυτό το μέσο και το Ταμείο ε, και τα υπόλοιπα ταμεία. Μετά, για τα θεματικ... τις θεματικές 1 και 2. Από τις πρώτες ε, προϋποθέσεις φαίνεται πως είναι πολύ πιο ψηλές οι προϋποθέσεις από ότι αυτές που είχαν συμφωνηθεί στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και μπορεί στην πράξη δηλαδή να είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ε, δύο λόγια για την ευελιξία και τη δυνατότητα ε, νέου προγραμματισμού. Αγωνιστήκαμε πολύ, πρόεδρος μαζί μας, ε, δεδομένου των τελευταίων υποθέσεων των φυσικών καταστροφών και σκέφτομαι το σεισμό στην Ιταλία. Αυτό το ποσοστό του 5% κατα... κατανομής υπό μία προτεραιότητα, πάντως όχι πάνω, όχι πάνω από το 30%. Ε, μπορεί να το ξαναδιαπραγματευτεί κανείς. Και έπειτα ρωτώ πάντοτε με στόχο να είναι όλα ε, χρήσιμα για τους πολίτες μας και για τις ε, περιφέρειες. Γίνεται μια αξιολόγηση για το πόσο αυτή η αλλαγή που έχει ήδη γίνει με το προηγούμενο Omnibus χρησιμοποιήθηκε, ήταν χρήσιμη ε, το χρησιμοποίησαν τα κράτη-μέλη και με τι τρόπο αυτή το... τον προγραμματισμό. Και κλείνω. Κλείνω με μια ανησυχία μου για τις ε, αποκαλούμενες ε, συνέργειες. Συμφωνούμε φυσικά για τις θετικές συνέργειες για το Horizon ας πούμε και το Seal of Excellence αλλά Υπάρχουν και πολλά προβλήματα και ρωτώ την Επιτροπή πώς σκοπεύει να λύσει, τη, να λύσει μάλλον να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τους οικονομικούς κινδύνους με συνεργείες για το Ταμείο Συνοχής Juncker 3,0. Αυτά είναι που μας ανησυχούν κάπως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο ακόμα Ομιλία Έχουμε δύο παρεμβάσει. Ο κύριος Μποστινάρου, παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο να είναι κανεί ε, σύντομο όταν έχουμε τόσο πολύ άριθμα προβλήματα και όχι λίγα. Και εδώ αναφέρομαι στο Ταμείο συνοχή. Χαιρετίζουμε το γεγονό ότι ε, το Ταμείο ERDF και το Ταμείο συνοχή βρίσκονται στον ίδιο κανονισμό. Και αυτό ακολουθεί και το πνεύμα τη δουλειά που κάναμε την περασμένη φορά, εγώ και ο Γιάνν Όλμπριχτ, τα δύο αυτά τα μία να γίνουν όχι ε, πλήρω ε, συμβατά, αλλά οι κανόνε είναι αρκετά κοντά. Στο Ταμείο Συνοχή όμω υπάρχουν κάποια πολύ ανησυχητικά ε, σημάδια. Πρώτον, τα κράτη-μέλη βλέπουν μια περικοπή 45% στο Ταμείο Συνοχής. Τεράστιο ποσοστό. Η Επιτροπή προτείνει να μεταβιβαστούν αρχικά 10 δισεκατομμύρια στην διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση. Τώρα στο τελευταίο σημείωμα αναφέρει 11,1. Και πρέπει να διευκρινιστεί και αυτό. Από πού προκύπτει αυτή η ε, διαφορά. Τρίτον, την προηγούμενη φορά καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα για την διευκόλυνση τη ιδιαίτερα στην Ευρώπη που μεταβιβάζονται από το Ταμείο ε, συνοχή θα μείνουν σε έναν ξεχωριστό φάκελο για μια τριετία. Διατηρείται τώρα η τριετία, αλλά ο εθνικό φάκελο μπορεί να ε, παρακρατήσει μόνο το 70% του συνδέοντα στην Ευρώπη. Δημιουργεί δύο προβλήματα αυτών. Ένα αρχικά σε εμά, στο Κοινοβούλιο, να διασφαλίσουμε την τριετία ε, στο πλαίσιο του ε, εθνικού φακέλου. Παράλληλα όμως ε, να διαγράψουμε την διάταξη που αναφέρεται στο 70%. Κάποια άλλα ζητήματα τώρα εν συντομία. Δεν υπάρχει ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμε πηγές ενέργεια στη στέγαση και επιλεξιμότητα των κλάδων αυτών υπό τους κανόνες όπως κάναμε την περασμένη φορά. Πρέπει να το διατηρήσουμε στην απρόταση. Καμία αναφορά στην, ε, στο 3Gen και στην ε, συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας γιατί αυτά είναι σημαντικά στοιχεία αν θέλουμε μια βιώσιμη οικονομία Μετά, ε, μείωση του συντελεστή ή αύξηση του συντελεστή σε χρηματοδότηση για το κράτος μέλος. Ήταν 85%, τώρα θέλουν 70% σε χρηματοδότηση. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό για τα κράτη-μέλη, εννοεί ο μιλητή. Στο παρελθόν είχαμε δει για τι φτωχέ περιφέρειε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα συγχρηματοδότηση Φανταστείτε τώρα που θα πάει στο 70% πόσο δύσκολο θα είναι. Μετά, υπάρχει μία αιμονή με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Κάτι στο οποίο έχει αντιταχθεί το Κοινοβούλιο. Και τέλος, προτιμώ να διατηρήσουμε τον ίδιο κανόνα 3 συν 1, αντί, μάλλον νη συν 3, διορθώνει ο μιλητής, αντί για τον νη 2. Και σας καλώ όλους να το σκεφτείτε γιατί δεν είναι το θέμα ποιο ε, ωφελείται και ποιος όχι. Τέλος, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι γίνεται να υιοθετηθούν οι ε, προτάσεις. Γιατί η Κομισιόν λέει ότι θέλει να υιοθετηθεί η Σύνοδος, ε, στη Σύνοδο μάλλον να υιοθετηθεί το όλο πλαίσιο και να διασφαλίσει και την υιοθέτηση. Με τις προτάσεις που μας παρουσιάσατε δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται με την μείωση της χρηματοδότησης και με όλα αυτά τα προσκόμματα πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να εργαστεί επί τούτου το επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ανοίξουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις ευθύνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε για τις ευκαιρίες που έχουμε να παραγάγουμε αποτελέσματα πριν τις ευρωεκλογές. Άλλο θέμα είναι αυτό. Και σίγουρα δεν είναι ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή συζητάμε μια πρόταση της Επιτροπής και εδώ αναφέρεστε στη δική μας ευθύνη. Στο μέλλον λοιπόν σας παρακαλώ να απευθύνετε ερωτήσει στην Επιτροπή διότι σήμερα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε απαντήσει. Και υπάρχουν και άλλες ερωτήσει, η κυρία Μάλετιτ. Αλλά σύντομα παρακαλώ αν θέλετε να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις έχω, όμως ε, θα κάνω μόνο μία πολύ σημαντική που έχει σχέση και με αυτά που ακούσαμε πριν ε, για τον ε, κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Ακούσαμε για την ενίσχυση των υστερούσων περιφερειών. Όμως τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων δεν κατάφερα να ε, βρω καμία αναφορά σε τοπικές ομάδες δράσης και οργανισμούς εκείνων των πολιτών κτλ. Δεν βλέπω λοιπόν κάποια τέτοια συμπερίληψη. Δεν βλέπω επίσης κάποια αναφορά στο Ταμείο ε, Γεωργικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι η προσέγγιση εδώ. Ε, με ποιο σκεπτικό πορευόμαστε. Επίσης, όταν ε, αναφέρεστε σε στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, τις οποίες βλέπουμε και όλες εδώ, και όταν αναφέρεστε σε στρατηγικές ε, εδαφικής ενοποίησης, ε, νομίζω πως υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός από την ευφυή εξειδίκευση και νομίζω πως αυτό είναι λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όλμπριχ, τώρα τελευταία ερώτηση. Ναι, ε, εγώ θα αναφερθώ στο κείμενο και όχι σε αυτά που ακούσαμε, διότι δεν ήμουν εδώ. Ε, διαβάζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέσα για την αστική ανάπτυξη. Από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια για ε, καινοτόμες αστικές δράσεις στις πόλεις. Εδώ τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα αποφασίσουν ε, τον διακυβερνητικό ή χαρακτήρα. Ε, αυτός όμως είναι ο τρόπος ε, να διαχειριστείτε εσείς το αστικό θεματολόγιο. Τι ακριβώ κάνετε. Η κυρία Βέστφαλ έκανε μια ερώτηση σχετικά με την αστική ανάπτυξη, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά που διαβάζω. Μπορείτε να μου τα εξηγήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φων Μπρέσκα, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Θα αρχίσω απαντώ στην ερώτηση του κυρίου Βαν Μίλτενμπουργκ, μια που δεν απάντησα στην προηγούμενη του ερώτηση για, το, ε, για τη σφραγίδα αριστεία και το πώς ε, θα λειτουργήσει όλο το σύστημα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά του κανόνε για τις κρατικέ ενισχύσει, θα μιλήσω με τεχνική γλώσσα εδώ, θα γίνει μια αναθεώρηση της, ε, του γενικού κανονισμού εξαιρέσεων αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε καθοδόν και αυτό τι σημαίνει ότι αυτά τα project με τη σφραγίδα αριστείας που θα χρηματοδοτούμε εμείς και όχι ο ορίζοντας θα ε, δέχονται την ίδια μεταχείριση σαν να χρηματοδοτούνταν από τον ορίζοντα. Θα, ε, τους, ε, θα διέπονται λοιπόν από τους ίδιους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. ο, κανονισμό μας, ο κανονισμός μας αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και όχι τις κρατικές ενισχύσεις. Χρειάζεται λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα έργα θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση ε, και χρηματοδότηση της Επιτροπής. Τι σημαίνει τώρα αυτό στην ουσία, στον κανονισμό μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτοματισμοί. Κάθε αρχή εξουσιοδότησης θα έχει την δυνατότητα να αποφασίζει αν θα χρηματοδοτεί κάποιο project ή όχι. Θα είναι λοιπόν στη δική τους ε, διακριτική ευχέρεια. Και μετά ε, ο διαχειριστής του εκάστοτε project θα μπορεί να πηγαίνει στην αρχή εξουσιοδότησης και να λέει «Να, ας πούμε, πήρα μια εξαιρετική πρόταση από την ε, Επιτροπή, νομίζω πως συμφωνεί με τους υπόλοιπους στόχους μας, τι λέτε». Και εάν υπάρχει συμφωνία, η αρχή εξουσιοδότηση θα λαμβάνει λοιπόν την απόφαση, η οποία, όπως είπα, δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, διότι θα διέπεται από άλλο καθεστώς, το οποίο ε, φυσικά θα ε, ρυθμιστεί από εμάς, από την Επιτροπή. Μετά, ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σίγουρα υπάρχουν συνδεσμένα μέσα στα ταμεία και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν γίνονται συζητήσεις για το πώς θα γίνονται αυτές οι συνδέσεις, διότι αυτή τη στιγμή οι συστάσεις είναι αναχώρα και όχι αναπεριφέρεια. Ε, γίνεται λοιπόν μια διαβούλευση ε, σχετικά με το πώς θα αλλάξουμε το επόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι και οι συστάσεις αναχώρα και οι γενικότερες εκθέσεις, εκθέσεις θα έχουν και κομμάτι για τις ε, επενδύσεις και ευρωπαϊκές και κρατικές οι οποίες όμως θα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση κάπως. Αυτό είναι δύσκολο λίγο να το προσαρμόσουμε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, όμως όπως σας είπα βρισκόμαστε σε στάδιο διαβούλευσης και αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε ένα δελτίο ε, ενημερωτικό για το πώς θα γίνει όλο αυτό. Δεν μπορώ βέβαια να μπω σε λεπτομέρειες γιατί όπως σας είπα βρισκόμαστε ακόμα σε στάδιο διαβούλευση. Ε, αστικές πρωτοβ... Ε, πρωτοβουλίες αστικής ανάπτυξης μάλλον. Τι γίνεται εδώ. Είχαμε 500 εκατομμύρια ευρώ στο 100... άρθρο 102 του κανονισμού. Μπορείτε να το βρείτε. είναι ο διάδοχος του Airbag, του Urban Innovative Actions και άλλων ε, πρωτοβουλειών. Προσπαθούμε λοιπόν να ενώσουμε όλες τις πρωτοβουλίες σε μία έτσι ώστε να προωθήσουμε ένα ενιαίο θεματολόγιο. Φυσικά δεν αντικαθίσταται ε, το υφιστάμενο πρόγραμμα ή μάλλον τα υφιστάμενα προγράμματα από τις νέες πρωτοβουλίες αυτές της Επιτροπής είναι κάτι που εστιάζει κυρίως στην ανταλλαγή γνώσεων και είναι πιο γενικό. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Βανίστελροι, ρωτήσατε αν περνάμε σε συγκεντρωτική, κεντρική διαχείριση. Ε, πρέπει πρώτα να, να απαντηθούν άλλα θέματα. Να πω ότι εμείς έχουμε ενισχύσει το ρόλο των ε, επιτροπών παρακολούθησης. Προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει οποιοδήποτε έργο, το σκεπτικό είναι ο ρόλος της να είναι ισχυρότερος ε, μέσω αυτής της Επιτροπής Ελέγχου. Για παράδειγμα τώρα υπάρχει υποχρέωση υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην Επιτροπή έτσι ώστε εμείς να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τον κατάλογο αυτό προτού επιλέξουμε ε, διάφορα έργα. Δεν αναφερόμαστε μόνο στα μεγάλα έργα, γενικότερα. Στόχος μας είναι να δούμε το πόσο υλοποιήσιμα είναι τα προγράμματα που προτείνονται. Δεν υπάρχει σίγουρα κανένας κίνδυνος ε, επιστροφής σε κεντρική διαχείριση. Έχουμε ενισχύσει το ρόλο τόσο της Επιτροπής όσο και ε, της ειδική Επιτροπής Παρακολούθησης. Τώρα, αστική ανάπτυξη. Να πω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Υπάρχουν απαιτήσει ε, για θεματική συγκέντρωση, για το περιβάλλον, για τις εκπομπές, ε, για την ε, χρήση λιγότερου άνθρακα. Το θέμα είναι που θέλουμε να φτάσουμε, διότι υπάρχουν και άλλοι τομείς που χρήζουν χρηματοδότησης. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε έστω και ελάχιστη ευελιξία στους υπεύθυνους διαχείρισης των προγραμμάτων, θα πρέπει, όπως λέει και η πρότασή μας, να υπάρχει κάποια ευελιξία, να υπάρχει αυτό το 6% δυνα... ως δυνατότητα μεταφοράς για να επέλθει ισορροπία. Ε, κύριε Μποστινάρου, να απαντήσω στα σχόλιά σας στο πλαίσιο του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζουμε τη στέγαση ιδίω των ε, πιο ευάλωτων ομάδων. Είναι εξάλλου ένας από τους στόχους πολιτικής μας. Το δεύτερο θέμα για την μεταφορά του 11,1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε άλλο ταμείο, να σας πω ότι αυτές είναι οι τιμές που έχουμε προς το παρόν. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής να επαναλάβω ότι όλο είναι θέμα επιλογών. Ή θα πεις ότι μας ενδιαφέρει η καινοτομία, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και αυτό θα στηρίξουμε, αλλά πρέπει να βρεις και τα ανάλογα χρήματα για να στηρίξεις όλα αυτά. Ε, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία για παράδειγμα, που τα ποσοστά είναι 12 ως 13% και όχι 33% όπως είναι στα νέα κρατημέλη. Υπάρχουν άλλες ανάγκες. Όμως αν έχει την άποψη ότι χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές στο περιβάλλον, τότε πρέπει φυσικά να κάνεις την επιλογή να διαγκώσεις το Ταμείο Συνοχής έτσι ώστε να μπορεί να, το, να καλύψει αυτές τις επενδύσεις. Δεν μπορείς όμως να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, όλα έχουν όρια. Σίγουρα αυτό μπορεί να συζητηθεί. Το γεγονός όμως ότι μειώνεται το Ταμείο Συνοχής δεν σημαίνει ότι οι πιστώσεις ε, κάποιου κράτους μέλους μειώνονται και αυτές με τη σειρά τους. Υπάρχει κάποια αναδιανομία ανάμεσα στα τρία ταμεία. Όμως, εάν η Επιτροπή σας, ε, για παράδειγμα, αποφασίσει ότι θέλουμε πιο πολλούς ε, δρόμους και λιγότερη εκπαίδευση, λιγότερες δεξιότητες, λιγότερη καινοτομία, τότε δυστυχώς πρέπει να επιστρέψουμε ε, στην κατάσταση που υπάρχει τώρα. Κύριε Ροπέ, αναφέρατε τον υπεθεματισμό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια έκκληση στα κράτη-μέλη να μην προσθέτουν κι άλλους κανόνες ε, σε αυτούς που ε, έχουμε ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ε, εξετάσουμε όλοι τις επιλογές απλούστευσης, ε, κόστους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει. Και τέλος. Νομίζω η κυρία Μάλιατιτς το ανέφερε. Γιατί όλες αυτές οι διατάξεις ε, τοπικής ανάπτυξης βρίσκονται ε, στον κανονισμό περί διατάξεων και χελού, γιατί απλά είναι διατάξεις οι οποίες ε, μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλα ταμεία, στο κοινωνικό ταμείο, ταμείο θάλασσας και ακόμα στο ταμείο ανάπτυξης της υπαίθρου, διότι υπάρχουν αναφορές στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εισαγάγαμε αυτές τις διατάξεις εκεί. Δεν συνεισφέρει μόνο ένα ταμείο στην ε, τοπική ανάπτυξη, αλλά πολλά. Είναι ένα σύνολο και το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου συνεισφέρει. Γι' αυτό λοιπόν ε, οι διατάξεις αυτές είναι στον, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και όχι στον κανονισμό για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Βανίσταν Ρόι. Είπατε ότι είναι πιο μικρή η πίτα και ούτω καθεξής. Γιατί όμως η ίδια μερίδα δίνεται στο ESF αφού γίνεται περικοπή στο Ταμείο Συνοχής. Το ποσό είναι το ίδιο με την προηγούμενη περίοδο. Αν έκανα τέτοια μοιρασιά στην οικογένειά μου, θα γινόταν χαμός. Ναι, κακώς αναφερθήκατε σε πίτες. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό παράδειγμα. Δεν έχω κάποια καλή απάντηση να σας δώσω σε αυτό το σημείο. Πράγματι, έχουμε ακριβώς το ίδιο ποσό τώρα με αυτό που είχαμε προτείνει το 14-20. 20 δις. Ε, συγγνώμη, 10 δις. Μπορείτε να πείτε ότι τα 10 δις στην προηγούμενη πραγματική περίοδο με βάση τις τιμές τότε είναι διαφορετικό ποσό σε σχέση με σήμερα. Με βάση τις σημερινές τιμές. Πράγματι λοιπόν είναι λίγο λιγότερο. Αλλά φαντάζεστε πόσο το συζητήσαμε αυτό το θέμα της μεταβίβασης και ποιο θα ήταν το ποσό και καταλήξαμε σε αυτό το συμβασμό στην Επιτροπή. Δεν έχω κάποια καλύτερη εξήγηση να σας δώσω. Γενικά, σαφώς και υπάρχει μια επανεξισορρόπηση στο πλαίσιο του προπολογισμού προς άλλες προτεραιότητες. Αλλά λυπάμαι δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα. Βλέπω ότι εδώ έχουμε τρεις από τους συντονιστές. Θεωρείτε ότι μπορούμε να αναστείλουμε την απογευματινή συνεδρίαση, γιατί έχουμε δύο ακόμα νομοθετικές προτάσεις μέχρι το 12.30. Το δέχονται οι συντονιστές. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Α, εννοείται την συνάντηση των συντονιστών. Αυτή να αναβληθεί. Στις 5. Εντάξει, συμφωνώ. Η κυρία Τόμας συμφωνεί. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με αυτή την πολύ σημαντική για μας συζήτηση. Ο κύριος Βαν έχει το λόγο για την επόμενη πρόταση. Interreg. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι σύντομος θα είμαι. Εδώ προτείνονται πραγματικά σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Όλα τα προγράμματα τα mainstream προγράμματα θα έχουν τη δυνατότητα της ε, προώθησης διαδικασιών και ενεργειών συνεργασίας μεταξύ περιφερειών. Δηλαδή, η συνεργασία δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του Interreg, αλλά και των κανονικών προγραμμάτων του ΣΥΡΜΟΥ. Ε, θα σας επισημάνω κάποια στοιχεία που εδώ αναφέρονται ως νέα. Το πρώτο που αλλάξαμε, και το είπα και προηγουμένως, είναι ότι έχουμε συγκεντρώσει τις νομικές διατάξεις που καλύπτουν τη συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά πλέον τα βρίσκεται στον κανονισμό ETC, που ελπίζουμε και πάλι να επιταχύνει και να απλουστεύσει την υλοποίηση. Εδώ τα κράτη-μέλη, τρίτες χώρες, χώρες εταιρικής σχέσης, όλοι έχουν ε, ίσα δικαιώματα ε, ψηφοφορίας, επιλογής ε, και συνεπιλογής των προγραμμάτων. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον ευνοϊκή διαχείριση προς τα κράτη-μέλη σε σχέση με, τις, με τους εταίρους μας. έχουμε, στη διασυνεργική συνεργασία έχουμε συμπεριλάβει και την, ε, και την θαλάσσια πολιτική, στην ε, υπερεθνική ή διεθνική συνεργασία για ε, τη θαλάσσια λεκάνη και τη σχετική στρατηγική θαλάσσιων λεκανών, ενώ παράλληλα επιτρέπουμε σε αυτά τα διμερή διασυνεργειακά προγράμματα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Μπαίνουμε λοιπόν περισσότερο στην ε, διεθνική συνεργασία του Ιντερεκ και δεν εντάσσονται τόσο στην ε, ε, διασυνοριακή συνεργασία. Αυτή είναι μια στρατηγική απόφαση για να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Όταν έχουμε πολλές περιφέρειες και χώρες που εργάζονται από κοινού σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη έχουμε ειδικό στοιχείο για τη συνεργασία των και απόκεντρων περιοχών, είτε μεταξύ τους είτε με, τους, ε, με τις γειτονικέ τους χώρες, για να οργανώσουμε τη συνεργασία και να τους δώσουμε περισσότερη ευελιξία και τέλος έχουμε και ένα νέο μηχανισμό διαπεριφερειακές επενδύσεις καινοτομίας. Εδώ θέλουμε να στηρίξουμε ε, και επενδύσεις και πιλωτικά έργα περιφερειών που προωθούν στρατηγικές ε, εφιούς εξειδίκευσης στους ίδιους τομείς προτεραιότητας. Στερίζουμε λοιπόν τις περιφέρειες ε, που εργάζονται σε έναν συγκεκριμένο ε, κλάδο σε όλη την Ευρώπη για την ίδια αλυσίδα αξιών. Θέλουμε λοιπόν να προαγάγουμε αυτές τις αλυσίδες αξίες και την ευφυή εξειδίκευση σε όλη την Ευρώπη τη διαχείριση αυτού του εργαλείου θα την έχει απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, προσπερνώ την επόμενη διαφάνεια. Περνώ κατευθείαν ε, στους στόχους πολιτικής. Ήδη τα ανέφερα προηγουμένως για το Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σαφώς και όλα αυτά ισχύουν και για το Ίντερεγ. Τρία όμως είναι τα σημαντικά στοιχεία για το Ίντερεγ. Πρώτον, και δεν αλλάζει αυτό, μπορούμε να καλύψουμε και δράσεις ε, τύπου ESF. Το ERDF λοιπόν μπορεί να πληρώσει αυτά που καλύπτει συνήθως το ESF. Δεύτερον, θέλουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε ε, την διαδικασία συμφιλίωσης ε, στην Ιρλανδία, στην ίσο της Ιρλανδίας. Οπότε υπάρχει μια σαφής τέτοια διάταξη για την προώθηση της ειρήνης και μετά το 2020 και μετά το Brexit. Μετά έχουμε μερικά στοιχεία τα οποία είναι ειδικά για το Interreg. Πριν από μερικού μήνε θα θυμάστε ότι υπήρξε ανακοίνωση τη Επιτροπή για τα ε, εμπόδια και προσκόμματα στα σύνορα νομική φύσεω. Με αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο πολιτική στηρίζουμε διασωνεριακές ε, περιφέρειες για την ε, αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Θα επανέλθω σε αυτό. Και μετά έχουμε και ένα στόχο πολιτική που συνδέεται με την ασφάλεια και την προστασία, ιδίω σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση των συνόρων, του μεταναστευτικού κτλ. Αυτή είναι η στόχη πολιτική που είναι ειδική για το Ίντερεκ. Και εδώ υπάρχει θεματική συγκέντρωση. Δεν ε, θα επισέλθω σε λεπτομέρειε. Απλώς να πω ότι για να έχουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση και όχι ad hoc σε συγκεκριμένα προγράμματα, κάποια κονδύλια τουλάχιστον θα πρέπει να διοχετεύονται σε συγκεκριμένο αριθμό ε, στόχων πολιτικής και για την αντιμετώπιση διοικητικών και νομικών προσκομμάτων και στενοπών στα σύνορα. Για τα υπερεθνικά προγράμματα ξέρετε ότι έχουμε μακροπεριφερειακές στρατηγικές που καλύπτουν 19 κράτη-μέλη, αν θυμάμαι καλά, και εδώ η πρόθεσή μας είναι κάθε μία από αυτές τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές να στηρίζονται και από ένα διεθνικό πρόγραμμα που να έχει ακριβώς ε, την ίδια εμβέλεια. Επόμενη διαφάνεια και πάλι χαμηλότερο συντελεστής σύγχρηματοδότηση 70% κατά κανόνα και για τα προγράμματα Interreg. Αλλά για τα εξωτερικά σύνορα νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε σε υψηλότερο ποσοστό, προτείνεται το 85%. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να τύχει μεγαλύτερη στήριξη σε αυτή τη συνεργασία, γιατί είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν σας παρουσιάζω αναλυτικά τα υπόλοιπα. Υπάρχουν κανόνες επιλεξιμότητας για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και έχουμε και σαφείς κανόνες για το Ταμείο Μικρών Έργων, Small Project Fund, το οποίο σαφώς θα πρέπει να τυχάνει διαχείριση σε ε, διασυνοριακού φορέα, και να υπάρχει συντονισμό για τα προγράμματα μέχρι ενός ε, ποσού, νομίζω 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία πλούστευση ισχύουν και για τα άλλα προγράμματα, ΦΠΑ, δεν υπάρχει προϋπόθεση για τα έργα ε, που παράγουν έσοδα. Υπάρχει όμως γενικά σημαντική μείωση του διοικητικού άκθου, Το τέταρτο σημείο για τους λογιστικού ελέγχου. Στην τρέχουσα πραγματική περίοδο κάθε πρόγραμμα Interreg ελέγχεται ε, μεμονωμένα. Στο μέλλον, επειδή για τα προγράμματα Interreg έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά σφάλματος, συνήθως κάτω από 2%, εδώ και πολλά χρόνια προτείνουμε να υπάρχει ένα δείγμα λογιστικού ελέγχου που θα καλύπτει όλα τα διασυνοριακά προγράμματα, αλλά με αυτό το δείγμα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ελέγχονται καθόλου και συνολικά το άχθος θα είναι πολύ μικρότερο. Αντί να κάνουμε λοιπόν επιμέρους ελέγχους ανά πρόγραμμα, θα έχουμε ένα μικρό δείγμα τυχαίο από πολλά προγράμματα. Γιατί βλέπουμε ότι λειτουργούν καλά τα προγράμματα Interreg. Και έτσι δεν χρειάζεται η συνήθις επαχθής διαδικασία λογιστικού ελέγχου. Αυτά. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν με τους ε, συντονιστές και τον εισηγητή. Θέλετε το λόγο? Όχι. Α, κυρία Ριμόντ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένο ότι, όπως είπατε και εσείς, το Interreg είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργούσε πάρα πολύ σωστά στο μέλλον και, κατά τη γνώμη μου, είναι ενδεικτικό της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και ε, των ευρωπαϊκών αξιών εν γέννη. Νομίζω πως ε, διαφημίζει ε, τη διασυνοριακή συνεργασία. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, το, ε, με την πρότασή της παρέχει στο Ιντερεγ ε, την κατάλληλη χρηματοδότηση. Το έχει εξοπλίσει με αρκετούς πόρους έτσι ώστε τα project που ε, στηρίζει να συνεχίζουν να δίνουν την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Θα ε, σας πάω στο άρθρο 7, 9. Ε, Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το σημείο 2 και γιατί ε, σημειώνεται ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση, ενώ αντίθετα μειώνεται στο 52,7% το σημείο 1. Πολύ σημαντική μείωση. Τι γίνεται λοιπόν με το ε, ε, Continuous Functional Areas, όπως λέει το πρόγραμμα στα αγγλικά. Τι σημαίνει αυτό. Στο άρθρο 16 μας είπατε κι εσείς ότι αναφέρονται οι επενδύσεις σε διαπεριφερειακά προγράμματα καινοτομίας, ε, παρότι το παρουσιάσατε, για να είμαι ειλικρινής, δεν το κατάλαβα και εντελώς. Αυτό που κατάλαβα από αυτά που είπατε είναι ότι το άρθρο 61 ορίζει ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι η αρχή διαχείρισης των ε, project αυτών. Για μένα ε, νομίζω πως όπως ακούσαμε και όλες οι χώρες, οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι υπεύθυνε για τη διαχείριση αυτών των διασυνοριακών project. Γι' αυτό λοιπόν και η ερώτησή μου αφορά τους στόχους τους οποίους έχει η Επιτροπή. Ποιος είναι ο σκοπός σας με ε, το να ορίσετε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την επιλογή των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν. Έπειτα, άρθρο 24, μικρά project, ε, project people to people και project για χρηστή διακυβέρνηση. Τι ακριβώ εννοείται με αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. κυρία Βέστφαλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. θα είναι αστείο γιατί παίρνω το λόγο για τη δική μου έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Νομίζω πως βάζουμε νερό στο κρασί μας και δεν χρηματοδοτούμε επαρκώς ε, τις ανάγκες μας. Η πολιτική συνοχή στο μέλλον χρειάζεται στήριξη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο τα διασυνοριακά κα μέτρα είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία, διότι αφορούν την καρδιά της Ευρώπης και χρειάζονται ακόμα περισσότερη χρηματοδότηση. Ακριβώς γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ε, είναι η διαφήμιση της προστιθέμενης αξίας της Ευρώπης. Η πρόταση λοιπόν προβλέπει τώρα λιγότερα κονδύλια, χαμηλότερη χρηματοδότηση για το Interreg και νομίζω πως χρειάζονται κάποιες εξηγήσεις. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Επίσης, εδώ θεωρώ προβληματικά τα ποσοστά χρηματοδότησης και εδώ έχω και κάποιες ερωτήσεις. Διότι όπως και ο Πασκάλ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ε, όλα όσα άκουσα. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερες ε, πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μικρά project. Πώς θα, χρημα... θα γίνει η χρηματοδότηση από αυτό το ταμείο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ τι θα συμβεί. Έπειτα, υπάρχει κάποιο παράδειγμα έτσι για να καταλάβουμε πώς ε, ακριβώς ε, θα ε, υλοποιηθούν αυτά τα διαπεριφερειακά, διασυνοριακά προγράμματα. Επειδή μπορεί να το κατάλαβαν άλλοι, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρη το έχω καταλάβει 100%. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόμασιτς, θα θέλατε το λόγο? Όχι. Κύριε Νταμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν για τον στόχο συνεργαφικής συνεργασίας ε, Interreg βλέπουμε να υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ισχυρό πλαίσιο και δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε χαμηλότερη ε, πρικοδότηση κατά 12%. 4 δις. 2,5% της ε, πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες περικοπές στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή να ησυχάσουμε ότι μόνο αυτό είναι. Και προστίθεται και η συνιστόσα για τις υπερπεριφερειακές ε, περιφέρειες, ε, τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες και για τα θέματα καινοτομίας. Ε, από ό,τι φαίνεται τα θαλάσσια διασυνοριακά προγράμματα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν και για το συγκεκριμένο ε, Έχουμε 28 προγράμματα διασυνοριακής θαλάσσιας συνεργασίας που βάζουν θεματικές πολύ σημαντικές για ολόκληρη την Ένωση. Ε, Αλλάζει ε, ανάπτυξη, ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός. Ακόμα και αν η Επιτροπή μας διαβεβαιώνει ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να συνεχιστούν, δεν διευκρινίζεται πώς ακριβώς θα συνεχιστούν μέσα σε αυτό το δεύτερο άξονα. έχουμε λοιπόν περισσότερο εντοπισμό σε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και σύμφωνο αλληλεγγύης. Θέλουμε δηλαδή οι εταίροι, οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δεύτερης συνιστώσας, όπου θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τις μακροπεριφερειακές ε, συνέργειες, αυτές κυρίως που αφορούν τις θαλάσσιες λεκάνες. Περισσότερη προσπάθεια ευελιξίας επίσης θα θέλαμε να υπάρχει και για τη συνέργεια τη θεματική για να αντιμετωπίσουμε ε, και τις περιφέρειες που ε, έχουν προσδοκίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάλετιτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ακούσω περισσότερα για αυτό το καινούργιο στοιχείο. Πώς ακριβώς ε, θα λειτουργεί στην πράξη. Γιατί χρειάζονται κανόνες σχετικά με την υλοποίηση, αλλά αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κανόνες για τις κρατικές ε, συμβάσεις Επίσης διαφέρουν και οι διαδικασίες από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Δεν είμαι σίγουρη λοιπόν πώς θα γίνει αυτό στην πράξη και τι θα απογίνουν τα project ε, τα οποία θα υλοποιούνται ανάμεσα σε ε, δύο χώρες IPA. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πρώτα να πω πως ε, συγκαταλέγομαι και εγώ στην ομάδα των ε, δυσαρεστημένων συναδέλφων, διότι αναμέναμε αύξηση της χρηματοδότησης της ε, δαφικής συνεργασίας διότι σε πολλά έγγραφα της Επιτροπής αναφέρεται ότι η αληθινή προστιθέμενη αξία βρίσκεται σε αυτά ακριβώς τα έργα και έχουμε μάλιστα πολλές περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών που αφορούν ακριβώς διαπεριφερειακά έργα συνεργασίας. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Κύριε Φανπρέσκα, είπατε ότι είναι δυνατόν η χρηματοδοτική οικονομική συνεργασία μπορεί να ε, στηρίξει διάφορα ταμεία. Μπορούμε λοιπόν να αντιλήσουμε ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για διάφορα project που αφορούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και ε, για το Ταμείο Θάλασσας. Υπάρχει η ναυτιλιακή συνεργασία, υπάρχουν διάφορες μορφές διακρατική συνεργασία, διάφορα προγράμματα. Μπορούμε να αναμένουμε το ίδιο και από το Ταμείο Θάλασσας και Ελίας, διότι μέχρι τώρα τα πάντα γίνονται στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε στήριξη από άλλα ταμεία. και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τόσο καλή συνεργασία ανάμεσα στα ταμεία στο παρόν πρόγραμμα της Επιτροπής. Αυτά είχα να ρωτήσω για το Interreg και σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω να δίνω κάποιες ε, απαντήσεις και μετά θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο που είναι ειδικό για τα θέματα που αφορούν το Interreg. Για να ξεκινήσω, όντως είναι αρκετά απογοητευτικό ότι το επίπεδο χρηματοδότησης δεν έχει αυξηθεί. Έχει μειωθεί όπως και ο ολόκληρος ο προπολογισμός και αυτό δεν είναι πολύ συνεπές και σύμφωνο με τις δηλώσεις που έχετε ακούσει. Είναι απογοητευτικό και ελπίζω πως θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου γιατί θα συμφωνείτε όλοι ότι έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία το ίντερ και θα πρέπει να στηριχθεί αυτό το πρόγραμμα και από οικονομικής άποψης. Το ερώτημά σας ε, ότι σε ποιο βαθμό το Κοινωνικό Ταμείο και το Θαλάσσιο Ταμείο μπορούν να συμβάλλουν. Ε, τα Interreg είναι προγράμματα ε, περιφερειακής συνεργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει πολύ, πολλαπλή χρηματοδότηση. Αν δούμε, ας πούμε, τις χώρες της Βαλτικής, θα... Εάν μιλάμε για τα κεντρικά προγράμματα που θα έχουν αυτές οι χώρες και τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης όπου ε, θα συγκεντρωθούν όλα αυτά τα κονδύλια, θα ήταν παράξενο αν έχουμε ένα κεντρικό πρόγραμμα δεν έχει αναφορά για το πώς, για το πώς σχετίζεται με τη συνεργασία ε, με τα υπόλοιπα τα Θα πρέπει να υπάρχει σαφή σύνδεση μεταξύ αυτού που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν και του πώς εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική συνεργασίας. Νομίζω πως εντασσονται στην ευρυτερη στρατηγικη συνεργασια νομιζω πως ειναι και υποχρέωση αυτό. Αλλά και πάλι δεν πρέπει αυτά να τα αναμειγνύουμε, να αυξήσουμε ας πούμε το Interreg ε, βγάζοντας δύο δις από το Ταμείο Συνοχής και πάλι πιστεύω πως μπορεί να γίνει αλλά ε, με διαφορετικό μάλλον τρόπο. Επίσης, τα χρήματα δεν χάνονται, απλώς έχει ληφθεί απόφαση να μετακινηθούν οι διασυνεριακές ε, συνεργασίες, μάλλον το διασυνεργειακό κομμάτι των θαλασσιών προγραμμάτων, γιατί έχουμε επίσης όχι μόνο χερσαία σύνορα, αλλά έχουμε και κάποια προγράμματα CBC που ε, αφορούν θαλάσσια σύνορα και έχουμε, θέλουμε να τα μεταφέρουμε στο ε, διεθνές κομμάτι του Interreg. Γιατί η ιδέα θα ήταν, ήταν ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο αν όλες οι δράσεις συνεργασίας, είτε είναι διασυνοριακού είτε διακρατικού τύπου, ε, ήταν κομμάτι της ίδιας, ε, του, ίδιου μάλλον στρατηγικού προγράμματος και προσέγγισης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο εταίροι που συνεργάστηκαν, ας πούμε η Ιταλία και η Κροατία, σε ένα πρόγραμμα CBC, ε, σε ένα θαλάσσιο σύνορο, ότι δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τέτοιου είδους διασυνοριακά προγράμματα. Όχι, μπορούν να συνεχίσουν. Επίσης λαμβάνουν τα ίδια ποσά, απλώς τα ποσά και το κομμάτι αυτό έχουν μετακινηθεί στο συστατικό 2. Δεν σημαίνει πως τα χρήματα χάνονται. Ήταν μια στρατηγική απόφαση. Τη Κομισιόν. Δύο λόγια ακόμα πριν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Έπρεπε να υπάρχει ε, συμβολή από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, το είπα, αλλά θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε και για το άλλο με ε, πλευρά των συνόρων. Θα είναι συμβολή, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες για το πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Άρθρο 61. Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην τεχνολογία και στην καιτονοτομία. Εάν να συνδυάσουμε όλες αυτές τις εταιρικές σχέσεις και στηρίξουμε την ε, δράση και πιο συγκεκριμένα να στηρίξουμε τις δραστηριότητε εμπορευματοποίησης. Και εδώ το πλεονέκτημα αυτό, εάν γίνει δηλαδή μέσω της Κομισιόν και δηλαδή αυτό σημαίνει βασικά υποβολή προτάσεων, πράγμα το οποίο θα ευθυγραμμιστεί με το πρόγραμμα Horizon, και πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες και τις κρατικές ενισχύσεις όπως εφαρμόζονται στο Horizon και αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία για να στηρίξουμε αυτές τις συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις. Dirk. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαριμών ε, ρώτησε για τις ε, contiguous areas. Εδώ πρόκειται για διεθνική συνεργασία στη θάλασσα, για μεγάλες περιοχές, ε, για διαπεριφερειακή συνεργασία. Για παράδειγμα, όπως ε, στην περίπτωση της ε, Φιλανδίας ή στο Αλκάρβα, στην Πορτογαλία. Τώρα, υπάρχουν ορισμένα αρκετά μάλλον μικρά project τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν. Και το People to People δημιουργήθηκε μετά από συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας στα σύνορα. Δημιουργήθηκε για να δημιουργήσει εμπιστοσύνη πρώτα ανάμεσα στους πολίτες ε, με ανταλλαγές μαθητών και ε, στη βάση αυτή σε έργα οικονομικά τα οποία θα μπορούσαν ας πούμε, να είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου το οποίο δεν έχει μεγάλο κόστος, λίγες χιλιάδες ευρώ. Στα ανατολικά σύνορα το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε ε, με διάφορους τρόπους. Στην Σαξονία, για παράδειγμα, στήριξε προγράμματα αξίας 200.000 ευρώ και το Ταμείο για τα μικρά project είναι ένα ταμείο που στηρίζει ακριβώς αυτά τα πολύ μικρά project και έχει και μικρό προϋπολογισμό. Στο Ταμείο λοιπόν για τα μικρά project μπορεί να υπάρχει ε, people του people, όμως ε, αυτό εξαρτάται από την περιοχή. Στη Λίμνη Κωνστάτσα, για παράδειγμα δεν ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που γίνεται είναι ότι καθίσταται σαφές ε, πως ε, στα πλαίσια του κανονισμού υπάρχουν συγκεκριμένες ε, λειτουργίες, συγκεκριμένα project τα οποία δεν διαχειρίζονται από μεσάζοντες, αλλά από τους δικαιούχους άμεσα. Και, για παράδειγμα, όταν διοργανώνεται ένα τουρνά ποδοσφαίρου ή ανταλλαγή μαθητών, αυτά είναι προγράμματα τα οποία υλοποιούνται άμεσα από τους δικαιούχους. Οι συμβάσεις που υπογράφονται δηλαδή είναι ε, άμεσες. Και οι τοπικές αρχές δεν ε, ασχολούνται με τη ε, διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, αλλά μόνο με τη γραφειοκρατία. Και να προσθέσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Φονπρέσκα για τα, το Μηχανισμό Προνταξιακής Βοήθειας και το CBC. Υπάρχουν τα προγράμματα ένδο Μηχανισμού Προνταξιακής Βοήθειας. Έμεση είναι η διαχείρισή τους και θα συνεχίσει να είναι έμεση. Η μεγάλη αλλαγή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στις χώρες ε, IPA είναι ότι ο κανονισμός αυτή τη στιγμή είναι εφιάλτης, υπάρχουν διάφορες ε, διασυνδέσεις, πολύ δύσκολο να τον ακολουθήσουμε ε, στην περίπτωση όμως αυτή θα ισχύει ο ε, απλός κανονισμός εκτός από συγκεκριμένα κεφάλαια εξωτερικής συνεργασίας για παράδειγμα και οτιδήποτε άλλο που αφορά ε, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ε, δημόσιες συμβάσεις θα ε, λαμβάνει χώρα κατόπιν συμφωνίας ανάμεσα στην ε, υποένταξη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Νομίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να ε, το συζητήσουμε πολλές φορές ακόμα. Ιδιαίτερα το ίντερνετ και τις ευκαιρίες που παρέχει. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με το τελευταίο θέμα, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, μηχανισμός επίλυσης διοικητικών διαφορών σε διασυνοριακό πλαίσιο. Η πρώτη πρόταση έγινε υπό Προεδρία Λουξεμβούργου. Τώρα έχουμε την πρόταση της Επιτροπής και ο κύριος Φονμπρέσκα θα μας την παρουσιάσει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, τι κρύβεται πίσω από αυτήν την πρόταση, ότι έγινε μια διασυνοριακή όριση ε, από το 2014 μέχρι το 2017. Έγινε, έγιναν κάποιες έρευνες, διαπιστώθηκαν διάφορες δυσκολίες στη συνεργασία, στη διασυνοριακή συνεργασία. Και ίσως θυμάστε ότι πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση όπου γινόταν απολογισμός της ε, διασυνορικής αναθεώρησης αυτής και βασισμένη σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι καλό θα ήταν να προτείνει ε, νομοθετικό κείμενο. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή ότι η νομοθετική αυτή πρόταση δεν έχει καμία σχέση με τον προπολογισμό ούτε με το Interreg. Επίσης, δεν πρέπει να συγχαίρεται με τις ε, υφιστάμενες ε, ομοδοποιήσεις εδαφική συνεργασία. Αυτή η πρόταση επιτρέπει δύο εταίρους που επιθυμούν να συνεργαστούν να χρησιμοποιήσουν τους ε, εθνικούς κανόνες του γειτονικού κράτους μέλους για τον σκοπό της ε, ομαλής συνεργασίας. Όπως είπα, για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ίσως το καλύτερο παράδειγμα που θα μπορούσα να σας δώσω είναι το τραμ ανάμεσα στο Στρασβούργο που το γνωρίζετε πολύ καλά και το Κέλ. Δείτε για παράδειγμα όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Χρειαστήκαμε 7 χρόνια από το μνημόνιο συνόησης μέχρι το ε, σύμφωνο για, ε, τους, ε, για τις χρεώσεις διότι υπήρχαν διάφορα διασυνοριακά θέματα, σήμανσης, ε, τιμολόγησης εισιτηρίων κτλ. Ήταν πολύ δύσκολο λοιπόν να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο και το σκεπτικό πίσω από την πρόταση είναι ότι αν είχαμε ένα εργαλείο που θα μας βοηθούσε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες θα επιταχύναμε την ε, υλοποίηση των ε, διασυνοριακών έργων. Δεν είναι όμως το Στρασβούργο το μόνο παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, συνεργατικής δραστηριότητας, στον τομέα της υγείας για παράδειγμα, ε, στον τομέα της ε, ασφάλειας. Αντιμετωπίζουμε στην, συνεχώς νομικές στενοπούς που μας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη και δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τα project με ταχύτητα που θέλουμε. Και θα περάσω στην τελευταία διαφάνεια. Βλέπουμε διάφορα νομικά μέσα τα οποία δεν έχουν καμία επίπτωση στον ε, κοινοτικό προπολογισμό. Δεν υπάρχει υποχρέωση χρήσης τους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ε, πρώτον, μέσω ανάληψης υποχρεώσεων, δηλαδή παίρνουμε από άλλο κράτος μέλος τα νομικά μέσα ή μέσω μιας δήλωσης που θα λέω ότι υπάρχει απέτηση για περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις από το εκάστοτε κράτος μέλος. Φυσικά, οι αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ε, τα οποία αφορά αυτή η διασυνοριακή συνεργασία. Δεν είναι απλά ε, δεν είναι τόσο απλό να χρησιμοποιήσει την νομοθεσία του γειτονικού κράτους μέλους. Πρέπει προηγουμένω να συμφωνήσουν οι αρμόδιε αρχέ του κράτους μέλους αυτού. Νομίζω πως αυτά είχα από μόνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις. Κύριε Βαν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιό. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή της. Παρότι νομίζω υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για την πρακτική εφαρμογή της. Επιλέξατε να εισαγάγετε ορισμό διασυνοριακής συνεργασίας στο επίπεδο ΝΑΤΣ 3. Ενώ ήδη έχετε αναφέρει αντίστοιχο μηχανισμό για την ε, αντιμετώπιση τέτοιων εμποδίων σε ό,τι αφορά ε, την υγειονομική περίθαλψη, υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Μπορείτε λοιπόν να το διευκρινίσετε αυτό το σημείο. Δεύτερον, η πρόταση θέλει να ε, δημιουργήσει διασυνοριακά σημεία συντονισμού, coordination points, χωρίς χρηματοδότηση όμως. Υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του ERDF υπό ε, προγράμματα περιφερειακής ή εθνικής συνεργασίας για να αυξήσει την οικοδόμηση δυναμικού και για αυτό το σκοπό. Γιατί θεωρώ ότι η χρηματοδότηση δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο ε, για τη θέσπιση αυτής της συνεργασίας. Επόμενο ερώτημα, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης, προβλέπεται λόγος, μόνο για, ρόλος μόνο για τα κράτη-μέλη, αλλά εφόσον πρόκειται για κανονισμό, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σωστή <clears throat> υλοποίηση αυτών των μέσων. Μετά, έχετε κατάλογο συγκεκριμένων παραδειγμάτων όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διασυνοριακό ε, μηχανισμό. Θίξατε το ενδιαφέρον παράδειγμα του Στρασβούργου, αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν μπει στο σιρτάρι αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια τέτοια διασυνοριακή συνεργασία. Κάποια στιγμή θα μπούμε και στον τριμερή διάλογο. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σα για την πρόταση των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μόρκοβα. ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την πρόταση της Επιτροπής, διότι λύνει πάρα πολλά διοικητικά θέματα στη συνοριακή συνεργασία και λύνει πολλά προβλήματα. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Μας δείχνουν ότι η κοινωνία είναι επιφορτισμένη με 60% περισσότερο διοικητικό κόστος για διάφορα διασυνοριακά έργα. Και εδώ προκύπτει και το πρόβλημα της ε, χρηματοδότησης της ε, διασυνοριακής συνεργασίας. Είπατε, αναφερθήκατε στο παράδειγμα της σύνδεσης με τραμ του Στρασβούργου και του Κέλ. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις εκτός από αυτή, για παράδειγμα ε, που σε περίπτωση πυρκαγιάς ε, έγινε κλίση στην πυροσβεστική του γειτονικού κράτους μέλους και δεν μπορούσε να περάσει τα σύνορα ακριβώ λόγω διοικητικού κολλήματο. Ε, ασθενοφόρα, μεταφορά ασθενών από μία χώρα στην άλλη, παρκαθυστερήσεις, ακριβώ λόγω αυτών ε, των ε, προβλημάτων συντονισμού σε διασυνοριακό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν η πρότασή σα να λύσει αυτά τα προβλήματα, να παραμερίσει τους φραγμούς που υπάρχουν και να ε, μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης. Βλέπουμε βέβαια θετικές ενδείξεις, όμως κανείς δεν ξέρει πώς ε, θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ε, πορεία. Τα κράτη τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν ή αν θα χρησιμοποιήσουν αυτά κέντρα συντονισμού ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος η πρόταση της Κομισιόν δημιουργεί έναν μηχανισμό ώστε τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τις ε, νομικές ε, ε, διατάξεις της χώρας εταίρου, αν υπάρχει αν υπάρχουν δηλαδή διαφορές. Εμείς θεωρούμε πως ο μηχανισμός αυτός ε, θα είναι προαιρετικός, δηλαδή ε, ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα συστήματα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η ρύθμιση όσον αφορά το σύστημα. Ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναλυθούν ε, ώστε να ε, εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του μέσου. Ποια είναι η λύση της Επιτροπής που προτείνεται γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Νταμάτο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, Όσον αφορά την ε, απλοποίηση και την ε, προσέγγιση της πολιτικής αυτής πιο κοντά στους πολίτες και λιγότερο βαριά από διοικητικής άποψης είναι ε, από ό,τι βλέπουμε αυτή η κατεύθυνση που ακολουθείτε. Ε, και το συζητήσαμε και στο Ιντερεγκ, αλλά επανεξετάζοντας σε επίπεδο διασυνοριακό, η Κομισιόν συνέλεξε στοιχεία πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με, τις με τα οποία οι συνοριακές παραμεθόριες μάλλον περιοχές έχουν χαμηλότερες επιδόσεις οικονομικές από άλλες περιφέρειες μέσα στα ίδια κρατή-μέλη. Οι δημόσιες υπηρεσίες όπως πανεπιστήμια ή νοσοκομεία είναι λιγότερο εύκολα ε, ε, και διαθέσιμα στις ε, περομεθόριες περιοχές και αυτό επίσης πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυφθούν μέτρα που θα ξεπερνούν τα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιοχές, γιατί στις παραμεθόριες περιοχές οι δυσκολίες δεν αντιμετωπίζονται μόνο μέσω Interreg. Ένας μηχανισμός για την εξάλληψη των νομικών ε, προβλημάτων ε, στις παραμεθόριες περιοχές είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα, όχι μόνο οικονομική στήριξη λοιπόν στο πλαίσιο του Interreg, αλλά και θεσμική στήριξη όπως οι ευρωπαϊκές ομάδες επιδαφικής συνεργασίας. Αυτές οι ομάδες, όπως γνωρίζουμε, ε, δεν έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες που θα μπορούσαν ωστόσο να επιτρέψουν να ξεπεραστούν τα νομικά ε, εμπόδια. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η προσφυγή σε αυτό το συγκεκριμένο μηχανισμό που γίνεται με βάση αυτό το μηχανισμό είναι θελοντικός, είναι προαιρετικός. Ε, μια χώρα μπορεί να αποφασίσει σε συνεργασία με κάθε όμορο κράτος να εξαλείψει τα νομικά εμπόδια. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους συνεργασία θα αποφασίσουν τα κράτη ε, μεταξύ τους, τα όμορα κράτη, είτε, αυτό, είναι, είτε είναι μέσα στην Ένωση είτε είναι εκτός. Περιμένουμε λοιπόν το σχέδιο του εισηγητή, αλλά λέμε από τώρα ότι θέλουμε να εστιάσουμε ειδικά στην οργάνωση αρμοδιοτήτων και σημεία συνεργασίας και συντονισμού για τις ε, διαμεθοριακές συνεργασίες, το ρόλο της Κομισιόν όσον αφορά αυτό το μηχανισμό και την νομική προστασία των ανθρώπων που διαμένουν σε διασυνοριακή περιοχή σε σχέση με τον ίδιο το μηχανισμό. Σας ευχαριστώ. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις όχι. Ο κύριος Φανμπρέσκα έχει το λόγο πάλι για να απαντήσει. Εδώ πρέπει να δώσω το λόγο στο συνάδελφο Ντέρκ. Μάλιστα. Όσον αφορά το οριοθέτηση της περιοχής, ΝΑΤΣ 3, πρέπει εδώ να είμαστε ειλικρινείς για αυτή την πρόταση. Η συγκέντρωση Μάλλον, η χρήση των εθνικών νόμων, της εθνικής νομοθεσίας ενός κράτους μέλους για να εφαρμοστούν και στην άλλη περιφέρεια του άλλου κράτους μέλους δημιουργεί ένα άλλο νέο νομικό όριο, σύνορο μάλλον, εντός αυτού του δεύτερου κράτους μέλους. Για να περιοριστεί αυτό ξεκινάμε λέγοντας ότι ε, πρέπει να μετακινηθούμε όσο γίνεται πιο κοντά στο, στα σύνορα όσο γίνεται. Ας πούμε για το τράμα ε, Εφόσον το τραμ ε, από το Στρασβούργο έχει το μεγαλύτερο του κομμάτι μέσα στο Στρασβούργο και μόνο τρεις στάσεις μέσα στο Κέλ, θα μπορούσε να ισχύσει για τις τρεις στάσεις εκεί, αλλά όχι για την, το υπόλοιπο, την υπόλοιπη πόλη του Κέλ και φυσικά όχι για ολόκληρο το κρατήριο της Βάδης Βουτεβέργης. Αν θέλουμε να διευρύνουμε το, το, το πεδίο, θα πρέπει να γίνουν σχετικές συζητήσεις, αλλά να αποφύγουμε τον κίνδυνο δημιουργίας νέων νομικών συνόρων εντός ενός κράτους μέλους. Το να χρησιμοποιηθούν ε, τώρα πιστώσεις από το Ταμείο Συνοχής ή από το Ίντερεγκ για να δημιουργηθούν σημεία συντονισμού, αυτό είναι δύσκολο γιατί... Ε, γιατί το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τέτοιου είδου κόστη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, οι περιφέρειες, επειδή είναι και στη συνθήκη, αλλά το Αναπτυξιακό Ταμείο θέλει να αναπτύξει κάτι και όχι να καλύψει λειτουργικά έξοδα, λειτουργικές δαπάνες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουμε. Η παρακολούθηση του σεβασμού και της στήριση των ισχυών των κανόνων δεν είναι θέμα της Κομισιόν. Φανταστείτε ας πούμε ότι για το τράμα αυτό η γαλλική νομοθεσία ισχύει ανάμεσα Γαλλία και Γερμανία, πρέπει κάποιος να παρακολουθεί αν τα βαγόνια του τραμ που κυκλοφορούν στη Γερμανία ε, τηρούν τους τεχνικούς κανόνες της Γαλλίας. Κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Είναι θέμα της Γαλλίας, είναι θέμα της Γερμανίας, ε, ο έλεγχος. Πάντως σίγουρα δεν είναι της Γερμανίας, ε, της Κομισιόν με συγχωρείτε, ο θέμα το να ελέγξει. Επίσης για την συνυπογραφή της δέσμευσης, για το αν δεν τηρείται, ε, όλα αυτά θα πρέπει να κοινοποιηθούν προς την Επιτροπή, ναι. Ο συντονισμός θα πρέπει να γίνεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Για νομικούς λόγους δεν μπορούμε αυτό να το βάλουμε στον κανονισμό, αλλά με βάση την, ανακοίνωση από το, του Σεπτεμβρίου για την συνοριακή συνεργασία, το συνοριακό ταμείο, ε, συγγνώμη, σημείο συντονισμού υπάρχει και αυτό κάνει ε, τον συντονισμό. Δεν έχουμε κατάλογο με παραδείγματα, αλλά θα ήθελα να σας παραπέμψω στην έκθεση ε, για τη διασυνορική συνεργασία, όπου έχουμε, έχουμε, μπορείτε να βρείτε μάλλον μια μακρά λίστα με νομικά εμπόδια, υπάρχουν και γλωσσικά εμπόδια, Η φραγμοί. Υπάρχει ένας κατάλογος λοιπόν, τον οποίο όμως δεν έχουμε τώρα εδώ μαζί. Τώρα, για την αντίδραση των κρατών μελών, δεν ξέρω τι μπορώ να πω για το Συμβούλιο, αλλά Η ομάδα εργασίας που έχει συνοδεύσει, έχει παρακολουθήσει την πρόταση της ε, ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου θα είναι η 8η ομάδα εργασίας ε, την επόμενη εβδομάδα και στη διάρκεια των 7 προηγούμενων συνεδριάσεων πάρα από 15 κράτη-μέλη συμμετείχαν και κανένας δεν είπε ότι δεν θέλει να το συνεχίσει. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα όσον αφορά την περιφερειακή ε, νομοθεσία και γι' αυτό και έχουμε φτιάξει αυτή τη διπλή προσέγγιση όπου το Σύνταγμα ενός κράτους μέλους δεν επιτρέπει ο Υπουργός να υπογράψει δέσμευση ε, βγαίνοντα από την κανονικά εφαρμοστέα νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένη εξαίρεση. Ωστόσο, όταν υπάρχει μια ανάληψη δέσμευσης, αυτό θα πρέπει να δημοσιευτεί στο, στην επίσημη εφημερίδα. Act adopted by the Parliament, there is a derogation for a limited uh, term τότε ε, αυτή αυτό μπορεί να ισχύσει λοιπόν για, για περιορισμένη ε, δαφική περιοχή. Για τον προαιρετικό χαρακτήρα, ναι είναι προαιρετικός, αλλά με την προϋπόθεση ότι αν το κράτος μέλος δεν επιλέξει τον μηχανισμό της Ένωσης, τότε υπάρχει ένας άλλος αποτελεσματικός μηχανισμός. Δηλαδή όταν το κράτος μέλος επιλέγει τον μηχανισμό, τότε βεβαίως είναι αυτό ολόκληρο το πακέτο. Έχουμε λοιπόν εκεί το περιφερειακό συντονισμό και τα περιφερειακά σημεία συντονισμού. Ε, αμοιβαία αναγνώριση, αλλά τότε δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο. Αυτός ο μηχανισμός δεν προτείνει αμοιβαία αναγνώριση, αλλά είναι ένα σύνολο κανόνων που ε, ισχύει και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Η αμοιβαία αναγνώριση είναι αυτό που όλοι βλέπουμε όταν ας πούμε παίρνουμε το δίπλωμα οδήγηση και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να νοικιάσουμε ε, αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι, αλλά δεν ισχύει αυτό για νέους οδηγούς ή για οδηγούς λεωφορείων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εάν υπήρχε αμοιβαία αναγνώριση, εντάξει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει για πολλά πράγματα, τότε ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει να εφαρμοστεί ένα σύνολο κανόνων. Επανέλθω στο παράδειγμα του ε, νοσοκομείου για να διευκρινίσω τη διαφορά στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Αμάτο και το, μηχαν... το μηχανισμό. Δηλαδή, το ίντερνετ είναι το μέσο. Δηλαδή, το, το νοσοκομείο μπορεί να φτιαχτεί από τη στήριξη του ίντερνετ. Όμως, το σώμα που διαχειρίζεται το νοσοκομείο είναι ACTC και η νομοθεσία δεν επιτρέπει να έχουν αυτή η ρυθμιστική αρμοδιότητα. Οπότε αντιμετωπίζουν πολλά νομικά εμπόδια, ιδιαίτερα για τους γιατρούς ή τις νοσοκόμες ε, που, εργάζονται στην Ισπανική, που είναι Γάλλοι και εργάζονται στην Ισπανία. Αλλά μέχρι στιγμής η Γαλλία έπρεπε να αποφασίζει για εξαιρέσεις. για να αποφασίζει πώς γίνεται όταν γεννιούνται στην Ισπανικά σύνορα, μάλλον στην Ισπανία τα παιδιά, τα βρέφη έχουν γαλλική εθνικότητα ή όχι. Έπειτα, κάτι που ε, διαπιστώσαμε από την εμπειρία μας όταν διαπραγματευόμασταν το κανονισμό ε, ε, GDC, δεν αφορά αυτό μόνο την προστασία των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή και άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε πάλι το παράδειγμα του τραμ. Μπορούν να πούν, ναι, ε, ε, έγινε ένα τύχημα και τραυματίστηκα γιατί δεν ίσχυε, δεν η νομοθεσία ε, που κανονικά ισχύει. Και αυτοί οι άνθρωποι προστατεύονται και ο κανονισμός λέει πού θα πρέπει να απευθυνθούν